Αξιότιμοι συνάδελφοι, καλωσορίσατε θερμά στη συνεδρία της Επιτροπής μας. Δευτέρα απόγευμα, αρχή μιας νέας εβδομάδας εργασίας. Σας καλωσορίζω ιδιαίτερα όλους. Σημείο πρώτο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Όπως βλέπετε, αύριο το πρωί δεν έχουμε ολομέλεια και θα μπορέσουμε να ε, διεξάγουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Γι' αυτό σήμερα αποσυμφορήσαμε λίγο την ημερήσια διάταξη και μεταθέσαμε θέματα για αύριο το πρωί. Δεν διαφωνεί κανείς από ό,τι βλέπω. Οπότε εγκρίνεται έτσι η ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Μπορώ να σας πω ότι στις 19 Ιανουαρίου η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων αποφάσισε με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να δηλώσουν τις μειώσεις τους, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στον ΟΗΕ και αποφασίστηκε να αναφερθούν και οι δύο αριθμοί 20% και 30% με δύο αστερίσκους. Γιατί το 20% ένας αστερίσκος που λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη ε, του, της Ένωσης δεν είναι μέλη εκεί και στο 30% τον άλλο γνωστό αστερίσκο ότι αυτό γίνεται δεσμευτικό από τη στιγμή που θα υπάρξει διεθνή συμφωνία με αντίστοιχες και συγκρίσιμες προσπάθειες ε, από πλευράς των εταίρων μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε σχέση με αυτό διαβάσαμε και ακούσαμε ότι Κάποιο ειπε είπε ότι 31η Ιανουαρίου δεν είναι, λέει, καταληκτική ημερομηνία, αλλά προσωρινή. Γιατί και στην Κοπεχάγη με εξέπληξε ότι αμέσω μετά τα Χριστούγεννα και αρχέ του χρόνου ε, προτάθηκε 31η Ιανουαρίου. Όλοι οι διαβοεί συμφώνησαν. Κανονικά θα θεωρούσε κανεί ότι ισχύει αυτή η ημερομηνία. τώρα λέει δεν ισχύει, δεν είναι καταληκτική και βεβαίω είναι αναμενόμενο ορισμένοι να καθυστερήσουν και να δώσουν τα στοιχεία εκπρόθεσμα, ελπίζω όχι πολύ αργά, στη Γραμματεία για την Προστασία του Κλίματος. Σε σχέση με αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Την περασμένη εβδομάδα έτσι έγινε μεγάλη φασαρία ε, στην Επιτροπή, στο πάνελ του IPCC για το ρυθμό με τον οποίο λιώνουν οι παγετώνες στα Ιμαλάια ε, αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπεται να ε, συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί σε μια συνεδρίαση και, μια έκθεση συνεδρίασης και συνέντευξη σε μια εφημερίδα ένα παγκόσμιο ε, επιστημονικό μάλιστα όργανο να καταλήγει σε μια διαπίστωση ε, η οποία δεν είναι έγκαιρη. Αυτό ρίχνει ε, νερό στο μήλο όλων εκείνων που αφισβητούν και τις επιστημονικές τεκμηριώσεις και τα στοιχεία για την κλιματική αλλαγή. Ζήτησε συγγνώμη τώρα το πάνελ για την κλιματική αλλαγή και έδωσε και εξηγήσει για το τι συνέβη, αλλά θα πρέπει να εκφράσουμε και εμείς κάποιες επικρίσεις. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα στη δική μας ε, ε, γνώση και αναγνώριση ότι είναι και ανθρωπογενής η κλιματική αλλαγή και υφίσταται προφανώς, αλλά δεν επιτρέπεται ε, να βγαίνουν τέτοια σε μια έκθεση και μετά ε, να περνάει από όλα τα Ινστιτούτα αυτά τα επιστημονικά και τα όργανα και σε ένα τόσο εξέχον όργανο να ισχυρίζεται κάτι. Κάποιος Ρώσος επιστήμονας είχε πει για το 2350 ότι θα λιώνανε και αυτό έγινε το 2035. Έγινε ο ρυθμός από 2350. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Το Κορεπέρ επίσης στις 19 Ιανουαρίου, όχι, λάθος, η Επιτροπή διορθώνει ο κ. Λάιν στις 19 του μηνός έκανε ανακοίνωση για τις επιλογές για μία ε, σύλληψη και ένα στόχο βιοπικιλότητας της Ένωσης για το διάστημα μετά το 2010. Αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει φέτος και ε, το έγγραφο το έχετε στη διάθεσή σας και εν ευθέτω χρόνο θα ε, συζητήσουμε και στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό. Και θα στείλουμε και αποστολή τον Οκτώβριο στη δεκάτη ε, διασκέψη στην Αγκόγια, στην Ιαπωνία. Αυτά ως ανακοινώσει του Προέδρου νομίζω και περνούμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 23ης Νοεμβρίου 2009 και 30ης Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα ε, θεωρηθεί εγκεκριμένο. Φτάσαμε ήδη λοιπόν στο σημείο 4. New impetus νέα όθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής, λέει, υδατοκαλλιέργειας. Η συγκήτρια είναι η κυρία Καρτίκα Λιωτάρ. Ε, Α, εδώ με βάλανε να κάτσω, γι' αυτό δεν με βλέπετε. Όλο και πιο αριστερά γλιστράς. Ε, Νόμιζα ναι, όσο αριστερότερα τόσο καλύτερα εδώ. Το λόγο έχει η συγκητρία. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Η έκθεση έπρεπε να είναι πολύ μικρή, πολύ περιορισμένη, κορσές, 1500 χαρακτήρες μου επέτρεπαν και εκεί έπρεπε να σταματήσω εγώ να περιοριστώ σε αυτό το πλαίσιο και βλέπουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερη παραγωγή και ζωική και φυτική, ε, ψάρια δηλαδή, αλλά και φυτική παραγωγή στις υδατοκαλλιέργειες και θα πρέπει να το δούμε με κάποιο κριτικό μάτι. Ε, προτείνω στην έκθεσή μου οπωσδήποτε η υδατοκαλλιέργεια να είναι και αηφόρος και δίκαιη από κοινωνικής πλευράς, δηλαδή ο κόσμος να μην εμποδίζεται συστηματικά ε, από τις βασικές του ανάγκες να έχει ε, πρόσβαση σε νερό, σε τρόφιμα και σε στέγη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές ε, στην Ινδία που διώχνουν αγρότες από την αγροτική γη και πλημμυρίζουν τα χωράφια για να κάνουν υδατοκαλλιέργειες, γαρίδες ας πούμε, προς εξαγωγή. Και ο κόσμος αποκτά και κοινωνικά προβλήματα και αυτό επηρεάζει κατά τα άλλα πάρα πολύ τη βιοπικιλότητα, διότι ε, κάνει και αλμυρό το έδαφος, και φάλμυρ, και Επίσης τα ψάρια είναι ζωντανοί οργανισμοί και πονάνε και στρεσάρονται και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Έχω κάνει δε και άλλες προτάσεις για να ε, μειωθούν ή να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δική μας επιτροπή, αυτό ε, ε, το εξετάζουμε και από πλευράς κοινωνικής, οικονομικής, βιοπικιλότητας και ευημερία των ζώων. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βλέπουμε ένα νέο φόρουμ για τις βιομηχανίες των βιολογικών προϊόντων και Έχουμε πολλά προβλήματα ήδη. Ε, θα πρέπει να εξάγουμε τα διδάγματά μας και να ε, ε, αποφύγουμε σφάλματα του παρελθόντος σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, τι προτείνω συγκεκριμένα. Να υπάρχει καλή ρύθμιση για να αποτραπούν να προληφθούν οι αρνητικοί συνέπειες, η ευημερία των ζώων επίσης να ληφθεί υπόψη σε μια αηφόρο υδατοκαλλιέργεια και να έχουμε μεθόδους αναισθησίας και μεθόδους θανάτωσης και μεθόδους μεταφορών των ψαριών με σύστημα πιστοποίησης αηφορίας. Και σε αυτό το σύστημα πέρα από την υγεία των ζώων θα πρέπει να κοιτάμε και το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, τα κοινωνικά στοιχεία, ε, τα οικονομικά, τα χρηματοπιστωτικά και προτείνω να λάβουμε υπόψη επίσης και να υπολογίσουμε στο γεγονός ότι η δατοκαλλιέργεια χρησιμοποιεί νέες μεθόδους ε, παραγωγής και θα πρέπει να μπει στον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, novel food. Και αν έχουν και άλλες καλές ιδέες οι συνάδελφοι, παρακαλώ να κάνουν τροπολογίες για να βελτιώσουν την πρόταση. Είπαμε 1500 χαρακτήρες δεν είναι πολύ κείμενο. Τουλάχιστον προσπάθησα τα σημαντικότερα να τα αναφέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Frau Kleiner Text, aber große Bedeutung. Μεγάλη σημασία ενός μικρού κειμένου. Σας ευχαριστούμε, κυρία Λιωτά. Άλλωστε η κατεύθυνση είναι όλο και περισσότερο προς ε, τεχνητή καλλιέργεια των ε, τροφικών αυτών ειδών. Έχουμε και άλλους που ζητούν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Ζέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε την εισηγήτρια. Σύντομη έκθεση αλλά πλούσια σε περιεχόμενο. Είναι αρκετά αρνητική η δομή της έκθεσης και μιλεί μόνο για προβλήματα του τομέα, ο οποίος τομέας ωστόσο έχει στο μεταξύ γίνει σημαντική πηγή ε, τροφίμων. Ίσως λοιπόν πρέπει να βάλουμε και κάποια θετικά πράγματα μέσα και όχι ε, να παρουσιάσουμε το όλο θέμα σαν δήθεν να είναι καθαρά αρνητικό. Γι' αυτό θα παρακαλέσω την εισηγήτρια να δεχτεί να περιλάβει ορισμένα θετικά. Για τη δική μας πολιτική ομάδα είναι σημαντικό τα ψάρια που παράγονται από τις ηχθειοκαλλιέργειες να είναι ασφαλή για τους καταναλωτές, βεβαίως με τήρηση των διατάξεων περί προστασίας των ζώων και εδώ έχει δίκιο η συγγέντρια είναι σημαντικό θέμα, αλλά βέβαια και η ασφάλεια των καταναλωτών πρέπει και αυτή να τονιστεί. Και χρειάζεται εδώ μια ίχνη λασιμότητα των παραγόμενων ψαριών. Από πού προέρχονται δηλαδή τα ψάρια που φτάνουν στην αγορά, όπως γίνεται και στο βόλιο κρέας. Αυτό θα προσφέρει και άλλη ασφάλεια. Όχι όμως μόνο μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, αυτό να αφορά και τα εισαγόμενα προϊόντα. Διότι εκεί ε, προκαλούνται σημαντικά προβλήματα από προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό το aqua labeling είναι κάτι το οποίο θα έχει θετικές επιπτώσεις. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα και το στοιχείο των περιβαλλοντικών συνθήκων για την καθιέρωση αυτού του eco-labeling. Τούτα θα βελτιώσουν στο σύνολο την κατάσταση. Σας ευχαριστώ, Ρίχα Τζέμπερ. Ακολουθεί ο Στρούαν Στίβενσον. Ευχαριστώ. Πρώτα, το ότι κάθομαι εδώ, κύριε Πρόεδρε, δεν σημαίνει ότι έχω αλλάξει πολιτικό προσανατολισμό με ευνηδίαζε. Χρειάστηκε να κοιτάξω ξανά και ξανά για να είμαι βέβαιο ότι είσαι εσύ. Καλά, ευχαριστώ τώρα την εισηγήτρια για τη σημαντική αυτή έκθεση. Θα κάνουμε και ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Αλία για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι στο προήμιο της έκθεσης η εισηγήτρια τονίζει πώς ε, ποιο είναι το μεγάλο δυναμικό των υδατοκαλλιεργιών. Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε στους εκτός ένωσης ανταγωνιστές μας να λάβουν πρωτοπόρο ρόλο. Πριν από 10 χρόνια εμείς ήμασταν η μεγαλύτερη παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες και επειδή σημειώθηκε μεγάλη αύξηση της ζήτησης για υγιή, υγιεινά μάλλον προϊόντα από ηχθειοκαλλιέργειες, πολλοί ρίχτηκαν για να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που έχουμε στην Ευρώπη, με, έχουμε ιδιώδες κλίμα, έχουμε ε, τεράστια ακτόγραμμη. Επιτρέψαμε όμως σε χώρες όπως την Χιλή, το Βιετνάμ, το Περού να μας ξεπεράσουν στην παραγωγή αυτή και να πλημμυρίσουν τις δικές μας αγορές με προϊόντα τα οποία πολύ συχνά είναι πολύ χαμηλότερων προδιαγραφών από αυτές που απαιτούμε να τηρούν η δική μας παραγωγή. Οι χτιοκαλλιεργητές στην Ευρώπη μου λένε ότι ο λόγος που σημειώθηκε αυτό είναι ότι γνωρίζουν ότι πριν να πουλήσουν έστω και ένα ψάρι πρέπει να σέβονται 400 διαφορετικούς κανονισμούς και όχι μόνο από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ αλλά και του εσωτερικού εμπορίου και του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Έχουν δηλαδή απέναντί τους ένα σωρό γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν. Έχουν τις κυβερνήσεις των χωρών μελών, έχουν, έχουν τις τοπικές αρχές και όλους τους σχετικούς ελέγχους που τους επιβάλλουν όλοι αυτοί. Τους κάνουμε τη ζωή αδύνατη δύσκολη πολύ εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο κλάδος αυτός παραγωγής ξεκίνησε από κάτι που θεωρούνταν κάποτε μη ασφαλές, βρώμικο, ότι προκαλούσε προβλήματα στο περιβάλλον. Έχει φτάσει όμως τώρα να είναι υγιεινή, καθαρή παραγωγή πρώτης ποιότητας, η οποία μάλιστα διασφαλίζει δεκάδες, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια της κοινότητας την ίδια στιγμή που οι αλληλευτικοί μας στόλοι μειώνονται. Άρα πρόκειται για κάτι που θα έπρεπε να το υποστηρίξουμε και να τους ανάψουμε όλα τα πράσινα φώτα σε εκθέσεις όπως της κυρίας Λιωτάρ. ...65.000 τόνους ενός ψαριού που λέγεται Παγκράσιους εισαγάγαμε από το Βιετνάμ. Πρόκειται για ένα ψάρι το οποίο ε, καλλιεργείται, ε, εκτρέφεται δηλαδή σε τεράστιες ε, θαλάσσιες φάρμες στο δέλτα του ποταμού Μεκόγκ και μεγάλες ποσότητες του ψαριού αυτού όχι μόνο εκτρέφεται αλλά και το επεξεργάζονται και μέσα στα νερά του ποταμιού αυτού που είναι από ό,τι έχουν δείξει διάφορα τεστ δύο ξύνες PCBs ακόμα και αρσενικό διάβασα κάπου ότι μερικά από τα ψάρια αυτά τους ε, βάζουν με ενέσεις ειδικέ ορμόνες που τις φέρνουν από την Κίνα με ε, στοιχεία από τα ούρα εγγύων γυναικών. Επειδή έχουν ορμόνες και το ψάρι έτσι θα αυξηθεί, δηλαδή το μέγεθος, το πάχος του ψαριού θα αυξηθεί και θα ε, οδηγηθεί ταχύτερα στην οριμότητα. 65.000 λοιπόν τόνους αυτού του ιδιαστικού ψαριού εισάγουμε στην Ευρώπη και <clears throat> πουλιέται στα σούπερ μάρκετ μας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ονόματα όπως ε, Panga Fish και Βιετναμέζικο Κόμπλερ για 2,5 ευρώ το κιλό κάνοντας την πραγματικότητα αληθινό dumping και undercutting οποιαδήποτε ε, τιμή που μπορούμε να ε, δώσουμε ε, στους αλείς ή στους ε, εμπόρους ψαριών όπου και αναλύονται αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει αρκετές, αρκετά, αρκετά τεστ από πλευράς κομισιών στα εργοστάσια αυτά του Βιετνάμ πριν να επιτρέψουν στο ε, Βιετνάμ. Ενώ υπάρχουν άλλα τέτοια ψάρια καλής ποιότητας από τις Φιλιππίνες που ε, εισάγονται επίσης, πάντως σίγουρα όχι από το Βιετνάμ. Εγώ νομίζω ότι η, Ευρωπαϊ... Ε, ότι η Επιτροπή μας θα προσφέρει πολύ μεγάλη υπηρεσία στις ευρωπαϊκές ηχθειοκαλλιέργειες αν στρέψει τα βλέμματά της και αρχίσει να εξετάζει τις πραγματικά αειδιαστικές αυτές εισαγωγές που φέρνουμε απ' έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ελέγχουμε λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, τους δικούς μας ηχθειοκαλλιεργητές οι οποίοι σέβονται τα τις υψηλότατες δυνατές προδιαγραφές για τις ε, παραγωγές που διοχετεύουν τις αγορές μας. Η έκκλησή μου λοιπόν προς τους συναδέλφους μου εδώ είναι να εφαρμόσουμε αυστηρές προδιαγραφές, αυστηρά πρότυπα σε όλες τις εισαγωγές και να δούμε πώς μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να ελαφρώσουμε λίγο τις ρυθμιστικές πιέσεις που εφαρμόζουμε στους δικούς μας ηχθειοκαλλιεργητές. Εγώ προτιμώ, εν πάση περιπτώσει, το φρέσκο ψάρι από τα νερά της Σκοτίας. Ο Κρήτον. Thank you very much, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δατοκαλλιέργεια είναι σημαντικό τομέα. Πρέπει να είναι μια δραστηριότητα αηφόρο και αυτό θα πρέπει να είναι ο σκοπό οποιοδήποτε κανονισμού. Οι προδιαγραφέ πρέπει να θεσπιστούν και για την παραγωγή μα και για τι εισαγωγέ. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή τη πρωτοβουλία πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση και έχει γίνει πολύ καλό έργο τώρα από τη συνάδελφο, την κυρία Λιωτάρ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία θέλω να δώσω έμφαση ωστόσο. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα της ασφάλειας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και των ζωοτροφών και των αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται για τα ψάρια. Είναι κάτι που δεν θεωρώ ότι έχει επαρκώς καλύψει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Γενικώς, ο κανονισμός που σχεδιάζεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρείται να επιφέρει διοικητικό άχθος. Όχι, δεν είναι έτσι. Το ζήτημα των αντιβιωτικών ε, και των ζωοτροφών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε και αυτή η δραστηριότητα να μπορέσει να είναι η φόρος. Επίτα η ανακοίνωση της Επιτροπής ακολουθεί μια κοινή προσέγγιση για όλα τα είδη δατοκαλλιέργειας, χωρίς διακρίσεις. Όμως υπάρχουν διαφορές μεταξύ πολυεθνικών ε, εταιριών και μικρών παραγωγών ή οικογενειακών επιχειρήσεων. Επίσης δίνεται έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες. Αυτά δεν φαίνεται ότι θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά περισσότερο τις πολυεθνικές. Και κυρίως για τα περιβαλλοντικά στοιχεία, Η ανακοίνωση της Επιτροπής ζητά έγγραφα για καθοδήγηση στον τομέα της θετοκαλλιέργειας, ιδίως στις περιοχές του Natura 2000. Και νομίζω ότι η θέση μας ως προς αυτό θα πρέπει να δώσει μεγάλο βάρος ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της ε, προστασίας της βιοποικιλότητας. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε κύριο Ντέιβις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 70% των ψαριών που καταναλώνουμε έχουν αλλιευτεί σε νερά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός αυτός είναι τόσο σημαντικός που δείχνει τη διαφορά μεταξύ ζήτηση και προσφορά στα ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν ξέρω πώ μπορεί οποιοδήποτε από εμά να μην παραδεχτεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί η υδατοκαλλιέργεια. Καλωσορίζουμε και το σχόλιο και την παρέμβαση του κυρίου Στίβενσον διότι μας δίνει κάποια περιστατωμένη γνώση για την υδατοκαλλιέργεια στην Σκοτία και δίνει και μια διαφορετική προοπτική των θεμάτων που μας απασχολούν. Εδώ ακούγονται πολλές τρομακτικές ιστορίες σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια εκτός Ευρώπης. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με νόσους των ψαριών, τα οποία εκτρέφονται σε δεξαμενές, όπως οι ψήρες. Επίσης η εκτεταμένη χρήση των αντιβιωτικών ή επίσης τα περιτώματα των ψαριών σε μεγάλες ποσότητες και η ρήπανση που μπορεί να προκαλέσουν στα ύδατα. Η διαφυγή των ψαριών και η ανάμεξή τους με τα ψάρια τα ελεύθερα και η δημιουργία μεικτών ε, κοπαδιών ψαριών και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα ζητήματα τα τονίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωση, όπω εγώ τουλάχιστον τα ερμηνεύω και τα διαβάζω. Η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να είναι υγιή, ασφαλή και να επιτρέπει και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού κλάδου. Και εγώ διαβάζω στι εφημερίδες ακόμη και στον τύπο τι τρομακτικέ αυτέ τι ιστορίε που σα έλεγα και πριν και όχι τι θετικέ πτυχέ που εμεί θέλουμε να τονίσουμε. Λοιπόν το θέμα είναι πόσο καλά τα πάμε στο να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Ε, το θέμα είναι από πού ξεκινήσαμε και ποιοι είναι οι σκοποί μας, τι επιδιώκουμε και πόσο καλά μπορούμε να συναγωνιστούμε χώρες εκτός Ευρώπης. Εδώ, αν κοιτάξουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής, ε, θίγονται κάποια ζητήματα βεβαίως, όπως αυτά που ανέφερε ο κ. Στίβενσον, όπως η υπόσχεση ότι θα πρέπει και τρίτε χώρε να σέβονται απαιτήσει τουλάχιστον ισοδύναμε με αυτέ που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει να ισχύει και για την εκτροφή των ψαριών τη υδατοκαλλιέργεια, αλλά και για την ποιότητα του κρέατος ψαριών που πωλείται. Ώστε να είναι σαφέ ότι δεν υπήρξε καμία απειλή ρήπανση, ότι μπορεί να πωλείται ε, ψάρι μολυσμένο από βαρέα μέταλλα που δεν ε, συμμορφώνονται με τους κανόνες ε, υγείας. Επίσης, με απασχολεί ένα ζήτημα που και αυτό θα ήθελα να θίγει κάπου. Μου λέγεται και ακούω συχνά ότι για να παράγουμε ένα, χιλιο, ένα ε, κιλό τόνου και ανοπτέρυγου τόνου χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ζωοτροφής για να παραχθεί αυτή η ποσότητα. Πολλές φορές η αναλογία είναι ένα προς τέσσερα και κάποιες φορές ένα προς ένα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ οι στόχοι μας να είναι λίγο πιο ξεκάθαροι. Να μας πει η Επιτροπή δηλαδή ποια είναι ακριβώς η κατάσταση σήμερα και πώς ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, λέγεται ότι θέλουμε να μειώσουμε τις εκφορτώσεις. Ε, αυτό πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο σύστημα για τις απορρίψεις. Ή επίσης το με τι είδους ψάρια θα ταΐζουμε άλλα είδη ψαριών. Υπάρχουν κάποια όρια σε αυτά. Διότι μπορεί να απειλήσουμε έτσι την ισορροπία της βιοπικιλότητας, ρηπαίνοντας ύδατα γύρω τουλάχιστον από τις περιοχές ε, των ε, υδατοκαλλιεργιών των ίδιων. Και επίσης να έχουμε και κατά νου τις ανάγκες των ε, καταναλωτών μας δεν μπορούμε απλώς να καλύπτουμε τις απαιτήσει των σούπερ μάρκετ εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τις συζητήσεις και να τις εξακολουθήσουμε σε επίπεδο επιτροπής, να επιδιώξουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους που φαίνεται όλοι να έχουμε από κοινού, δηλαδή να προωθηθεί η δατοκαλλιέργεια, αλλά ασφαλής, υγιής και να είναι και επιχειρηματικά βιώσιμη. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντέβης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές οι προκλήσεις και ε, ο κλάδος είναι ταχαίως αυξανόμενος και καλή έκθεση. Ε, μια λεπτομέρεια για το σημείο α ίσως, όπου γίνεται για αναφορά σε ένα κατάλογο προβλημάτων ενδεχομένων. Βεβαίως ε, περιλαμβάνει και το διοξίδιο του άρθρακα, το οποίο όμως είναι λίπασμα που χρειάζονται τα υδρόβια φυτά. Και κάτι άλλο. Και κάποια χημικά που βλέπουμε στον ΟΠΟ ε, στο γλυκό νερό PCB και ιστρογόνα που συνδέονται με το φύλλο και με τα ψάρια και με τους ανθρώπους. Αυτά δεν είναι υποπροϊόντα των υδατοκαλλιεργιών, αλλά τα επηρεάζουν και τα ε, προϊόντα τους. Στη Βρετανία γίνονται ε, μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα για ερμαφρόδιτα ψάρια που παράγουν και τέτοιες ουσίες και χημικές και επηρεάζουν και το ανθρώπινο σύστημα αναπαραγωγής και έχουμε ε, διαμαρτίες ε, στη γέννηση και προβλήματα άλλα και κλονίζεται και η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη σε ένα πολύ σημαντικό κλάδο της ε, βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Η Εστέρ Δελάνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αφού ήρθε ο Πολ κάτι να μας εξηγεί τη Δευτέρα ότι δεν θα πρέπει να τρώμε κρέας, Αφού τα ακούμε όλα αυτά, δεν ξέρω αν έχουμε όρεξη να τρώμε και ψάρι. Ε, είναι όμως σημαντικό ε, να σημειώσουμε την πρόταση που έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι ότι η υδατοκαλλιέργεια αυτή καθ' αυτή δεν είναι προβληματική, δεν είναι κακή. Η έκθεση ε, επικεντρώνεται πολύ στις ανετικές συνέπειες. Πόσο ήταν, 1500 χαρακτήρες είπατε. Εντάξει, ένα κείμενο όμως που λέει ότι καταρχήν δεν υπάρχει πρόβλημα με την υδατοκαλλιέργεια, αλλά ε, το θέμα είναι τι ε, τρόφιμα θα παράγουμε με τρόπο ελεγμένο, με λιγότερο παρεμβατικές και επιθετικές μεθόδους για το περιβάλλον και για ε, τον άνθρωπο από ότι η Αλία. συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνει. Έχω δύο προτάσεις. γιατί επικαρτικά κάντε τροπολογίες, γιατί εγώ δεν έχω ε, πολλές λέξεις παρά μόνο 1500 χαρακτήρες. Εγώ έχω να προτείνω δύο πράγματα. Το ένα το είπε και ο Στίβενσον. Ε, πρόσφατα ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι πρόθυμη να κάνει έρευνα για τον τρόπο παραγωγής και τις μεθόδους παραγωγής σε συγκεκριμένες ε, ασιατικές χώρες, τη λάπια ή ε, παγράσι φιλέτα, πώς παράγονται εκεί και στο Βιετνάμ και σε άλλες χώρες και με βαρέα μέταλλα που υπάρχουν στο νερό και περνάνε και στα ψάρια και ρώτησα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κινδύνους στη δημόσια υγεία γιατί αυτό είναι ο δικός μας ρόλος, της δικής μας Επιτροπής. Θα κάνω λοιπόν πρόταση, παρακαλώ να το κοιτάξει η καρτίκα για να απευθύνουμε από κοινού την έκκληση αυτή. Και ένα δεύτερον, τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα παγκοσμίω σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τις μεγάλες διαφορές στην νομοθεσία. Έχουμε μεγάλες εταιρείε παραγωγής ε, και ευρωπαϊκές που πάνε, ξέρω εγώ, στη Χιλή, γιατί είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές και απαιτήσει χαμηλότερες. Θα πρέπει να καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να λέμε ότι τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν ε, ανταποκρίνονται στις ίδιες προδιαγραφές, τα ίδια πρότυπα, δεν θα πρέπει να παίρνουν άδεια να κυκλοφορούν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να ξεφορτωθούμε αυτά τα προβλήματα. Συγκεκριμένε προτάσει για τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ, Εδώ τέθηκαν πολλά σοβαρά ζητήματα και πολλές ερωτήσεις εύστοχες ήδη έχουν τεθεί. Θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους ήδη για τα όσα είπαν. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω λοιπόν εδώ ένα δικό μου σχόλιο Υπάρχουν πληροφορίες για το πόσος χώρος απαιτείται από, για κάθε είδος ψαριού στα πλαίσια της υδατοκαλλιέργειας και βάσει των συστημάτων που εδώ προτείνονται, διότι ακούμε ότι τα ψάρια υποφέρουν και αυτά από πόνο και άγχος και στρες. Και αυτό μπορεί να οδηγεί στην παραγωγή ορμονών που να βλάπτει την ποιότητα του κρέατος. Επίσης ακούσαμε για τη χρήση των αντιβιωτικών των ε, ορμονών στα ψάρια και αυτό μπορεί τελικά να καταλήγει σε εμά, στο δικό μα οργανισμό όταν καταναλώνουμε κρέα ψαριού. Τι, γεγονός, τι στοιχεία λοιπόν έχουμε για το χώρο που διατίθεται στις, ε, στην εκτροφή ψαριών στι υδατοκαλλιέργειε. Πόσο χώρο χρειάζονται τα ψάρια ανάλογα με το είδο του ώστε να μην υποφέρουν από στρε. κύριος Σκυλακάκης, παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικά σχόλια. Πρώτον, με ποιο τρόπο και γιατί δίνει η έκθεση αυτή την εντύπωση ε, για το υδατοκαλλιέργειες αν είναι καλό ε, ή κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποια επιφύλαξη. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου υπάρχει εδώ μια βασική αρχή που δεν αναφέρεται στην έκθεση και είναι η εξής. Η υδατοκαλλιέργεια μας επιτρέπει ουσιαστικά να προστατεύουμε και να διαφυλάσσουμε μέρη του περιβάλλοντος που επιβαρύνονται ιδιαίτερα από την υπεραλίευση. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο ολόκληρο. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι απειλές και οι πραγματικοί κίνδυνοι της υπεραλίευσης και είναι και παγκόσμιοι. Αυτό το σημείο νομίζω θα πρέπει να μπει στην έκθεση. Δηλαδή, να μην λέμε απλώς ότι εντάξει είναι ακόμα ένας κλάδος. Όχι, έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν γίνεται με σωστό τρόπο. Ένα αυτό σχόλιο. Παρατήρηση δεύτερη τώρα. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους ε, που αναφέρθηκαν στον αθέμητο ανταγωνισμό και σε ορούς περιβαλλοντικούς αλλά και σε ό,τι αφορά τις προφυλάξεις για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε αυτό το στοιχείο και να το αναφέρουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα απολύτως. Αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι για το θέμα της ατοκαλλιέργειας έχουμε να κάνουμε με μια πτυχή της βιώσιμης ανάπτυξης εδώ, που μας δείχνει ότι σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Η υδατοκαλλιέργεια από τι προκύπτει, η ανάγκη της υδατοκαλλιέργειας μάλλον, από τις συγκεκριμένες ανάγκες ειδών ψαριών και από τον κίνδυνο εξαφάνισής τους. Και βεβαίως με ανάλογη επίδραση και στην ισορροπία της διατροφής. Έτσι λοιπόν η έμφαση στην υδατοκαλλιέργεια πρέπει να δοθεί ανάλογα με το τι χρησιμοποιεί για να για να τρέφει αυτά τα ψάρια και ξέρουμε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται μικρότερα είδη για τα μεγαλύτερα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς θα μπορέσουμε στα πλαίσια αυτής της τάξης να έχουμε μια κοινή, μια σφαιρική προσέγγιση του όλου θέματος. Ευχαριστώ εδώ την συγκεκριά μας για τα διάφορα ζητήματα τα οποία φώτισε με τη σύνταξη της έκθεσής της, όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας, περιεχομένου, ένα θεωρητικό ζήτημα. Όποτε ενσκέπτουμε σε ένα περιβαλλοντικό θέμα, κυρίως ω προ τη διάθεση των πόρων, δεν θα πρέπει να προκρίνουμε λύσει που να προκαλούν τελικά νέε δυσκολίε. Θα πρέπει δηλαδή να σταθμίζουμε προηγουμένω τι συνέπειε. Μην ε, θεραπεύουμε ένα πρόβλημα με ένα καινούριο. Άρα εδώ αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς η δατοκαλλιέργεια θα είναι αηφόρο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση για τα διάφορα είδη ψαριών που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια και πώ δεν θα μετατοπιστεί το πρόβλημα αλλού βεβαίω, διότι έτσι δεν επιλύουμε κανένα θέμα. Έτσι λοιπόν η παρέμβασή μου δεν περιέχει ερώτηση, ούτε προτείνει κάποια απάντηση, αλλά θα έλεγα εδώ να σκεφτούμε κάπως μεθοδολογικά το θέμα. Δηλαδή, ως προς την ευαντοκαλλιέργεια, βρισκόμαστε και πάλι ενώπιον ενό προβλήματο που είναι ένα πρόβλημα γενικό, ευρύτερο, το οποίο θα μας απασχολεί κάθε φορά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη συρρήκνωση των διαθέσιμων πόρων. Των πόρων που έχει στη διάθεσή τη η ανθρωπότητα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, τι μελέτη αντικτύπου θα έπρεπε να προβλέψουμε για τις, προτινόμενε για τις προτινόμενες λύσεις, επιλογές που... μεταξύ των οποίων θα πρέπει να διαλέξουμε και να φροντίσουμε η απόφαση που θα... Ε, στην οποία θα καταλήξουμε να μην είναι χειρότερη από την κατάσταση που ήδη ισχύει. Ευχαριστώ. Πρόσφατα συμμετείχα σε, ένα συνέδριο για υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή μου και έμαθα ότι οι περισσότεροι τόποι όπου υπήρχαν υδατοκαλλιέργειες έκλεισαν διότι δεν τα κατάφερναν καλά αυτοί που τις λειτουργούσαν. Συχνά λοιπόν είχαν αποτυχίες λόγω νόσων, λόγω μόλυνσης, λόγω νόσων των ψαριών και ούτω καθεξής. Κάτι που δείχνει ότι πολλοί ρίχτηκαν στην επιχείρηση αυτή για να βγάλουν γρήγορα λεφτά και στην πραγματικότητα δεν είχαν ενημερωθεί καλά, δεν τα ξέρανε καλά, ενώ και επιστήμη αυτή. Το αποτέλεσμα είναι ότι εκατομμύρια τόνοι ψαριών χάθηκαν με τον τρόπο αυτό, γιατί όπως είπα, για να γίνει η θεοκαλλιέργεια σε εσωτερικά ύδατα, λίμνες και τέτοια, χρειάζεται όπως είπα πολύ βαθιά γνώση. Τώρα είχαμε ερωτήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ποιοτικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους ελέγχους των εισαγωγών. Θα μας ενημερώσει σχετικά ο κύριος Βάισεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να θυμίσω το πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής. Και ακούμε εδώ περίπου αυτά που έχουμε συζητήσει με τους διάφορους ενδιαφερομένους του κλάδου τα τελευταία δύο χρόνια. Ξεκινήσαμε από μια διαπίστωση και το είπαν πολλοί εδώ. Γενικά η δατοκαλλιέργεια είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται ταχύτατα ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό στον κόσμο γιατί αυξάνεται και η ζήτηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ευθύ εξ αρχής γιατί έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια. Όταν μιλάμε για υδατοκαλλιέργεια πρόκειται για όλους τους ζωντανούς υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να είναι ζώα, μπορεί να είναι φυτά, αλλά και για την Ευρώπη για ζώα δεν είναι μόνο τα ψάρια, είναι και τα οστρακοειδή. Και ε, τα οστρακοειδή είναι το ίμιση και πλέον της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτή τη στιγμή. Επανέρχομαι στο πλαίσιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τη διαπίστωση που λέει ότι όντως μετά από μια στρατηγή για η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας το 2002 έγιναν τεράστιες πρόοδοι από πλευράς περιβαλλοντικής αηφορίας. Επίσης, απόλυτα σεβόμαστε ε, τους ε, κανονισμούς υγιεινής και για την προστασία των καταναλωτών αλλά και για την προστασία των ζώων των ίδιων. Ωστόσο, τα τελευταία δέκα χρόνια διαπιστώσαμε ότι η συνολική παραγωγή ε, των υδατοκαλλιεριών στην Ευρώπη δεν έχει μεταβληθεί. Δηλαδή, 1,2-1,3 εκατομμύρια τόνοι περίπου είναι η ευρωπαϊκή παραγωγή και παραμένει αυτή σταθερή. Ενώ περιμέναμε σημαντική αύξηση ε, της παραγωγής αυτής. Συνεπώς, από το 2000 και μετά ξεκινήσαμε με ευρύτατη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών για να δούμε ποιοι είναι αντικειμενικοί λόγοι αυτής της αποτελμάτωσης. Ήταν απλή σχετικά η διαπίστωση. Σε γενικές γραμμές υπάρχει συνένεση για να πούμε ότι η Ευρώπη ενδεχομένως να ε, εφαρμόζει τους πιο αυστηρούς όρους και προδιαγραφές για την προστασία και του περιβάλλοντος αλλά και του καταναλωτού. Παράδειγμα, και μετά τη στρατηγική του 2002 εγκρίναμε έναν κανονισμό ο οποίος ελέγχει την εισαγωγή ε, μη ε, ε, ηθαγενών οργανισμών που ονομάζονται εξωτικοί οργανισμοί στις υδατοκαλλιέργειες για, να, για την προστασία της βιοπικιλότητας και την αηφορία. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω και να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε η υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσεται στην Ευρώπη να, μην είναι αηφόρος από πλευράς περιβαλλοντικής. Έτσι λοιπόν και προς το σκοπό αυτό τονίστηκε μια σημαντική πρόκληση και από τον κύριο Στίβενσον και αυτό είναι ο αριθμός των νομοθεσιών, των, νόμων, όχι μόνο ε, της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και της εθνικής. Και από την άλλη ε, δεν υπάρχει ε, θεμητός ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες. Δηλαδή ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται από τα προϊόντα που εισάγουμε. Επίσης γνωρίζετε, όπως εγώ, ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα ως προς την ασφάλεια του καταναλωτού ε, που θα πρέπει να ε, φάγονται στους ίδιους κανόνες, στους ίδιους νόμους ή στην αντιστοιχεία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όμως ότι η εξοκοινωτική παραγωγή δεν έχει τους ίδιους κανόνες και πρότυπα για το περιβάλλον και την προστασία του καταναλωτού και είναι πολύ δεινή η θέση μας. Έχουμε αιτήματα λοιπόν για ισότητα. Εμείς συνεχίζουμε να προωθούμε την ασφάλεια των τροφίμων, βέβαια θα γίνει αλλού η συζήτηση αυτή, για να υπάρχει μια ευρύτερη ε, παγκόσμια διακυβέρνηση και για τα προϊόντα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσω συγκεκριμένα σε κάποιο σημείο της συζήτησης, γιατί εδώ ε, ακούστηκαν και θέματα διατροφής και θέματα ε, αντικτύπου περιβαλλοντικού και ρήπανσης ο κανονισμός novel food, η κλωνοποίηση που αναφέρεται και στο σχέδιο της Ήτριας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ähm, ich sehe, Τέθησαν ερωτήσεις. Ο Κρίς Ντέιβις όμως έχει συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκρίνηση που έδωσε. Αλλά στο έγγραφό τους, στο έγγραφό της Επιτροπή δηλαδή, λέει ότι σχετικά με την ευημερία των ζώων και την προστασία του καταναλωτού θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ε, χώρες από τις οποίες γίνονται εισαγωγές τηρούν πρότυπα, προδιαγραφές, τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που τηρούν η ε, Ευρωπαίοι παραγωγοί. Και τώρα μόλις είπατε δεν μπορείτε να το κάνετε. Τι γίνεται τώρα, ίσως αυτό το βρετανικό σύστημα marine stewardship που εγγυάται ότι τα ε, ψάρια και άλλα προϊόντα θάλασσας ε, σέβονται ορισμένα πρότυπα ε, μπορεί να επεκταθεί. Αλλά τι θα κάνετε πιο συγκεκριμένα. Ναι, αυτό ρώτησα κι εγώ. Ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια διάκριση. μια είναι η δημόσια υγεία και από την άλλη το περιβάλλον, η ευμερία των ζώων κτλ. Και εγώ γνωρίζω καλά την νομοθεσία και είναι πιο εύκολο να αφήσει ένα προϊόν έξω από τις θύρες της Ευρώπης όταν απειλεί τη δημόσια υγεία παρά όταν απειλεί άλλα πράγματα. Ωραία, ας πάρουμε τη δημόσια υγεία τώρα και μόνο. Ε, αφού έχουμε ένα εργαλείο για να αφήσουμε έξω ακριβώς τα εξωτερικά προϊόντα εφόσον υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει επανειλημμένα ότι «Α, ναι, για τη δημόσια υγεία βεβαίω θα πρέπει να τηρούν τι ίδιε προδιαγραφέ και του ίδιου όρου με τα ευρωπαϊκά προϊόντα». Μα εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό πώ θα το ελέγξετε παρακαλώ. Με τον ίδιο τρόπο τη βιολογική παραγωγή στην Κίνα α πούμε. Δηλαδή περιμένετε να σα στείλει ένα φάξ που να λένε οι Κινέζοι ότι τα προϊόντα αυτά είναι βιολογικά. Το πιστοποιούμε αυτό θα κάνετε ή θα πάτε επί τόπου να δείτε πώς παράγονται αυτά τα περίφημα βιολογικά προϊόντα. Και δεύτερη ερώτηση και γραπτή ερώτηση έχω υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένω τέσσερις εβδομάδε να μεταφραστεί και να μου απαντήσετε. Ωραία να δω αυτά που θα μου απαντήσετε τι θα είναι. Και είστε πρόθυμοι να κάνετε αυτή την έρευνα. Ποιοι είναι ε, η παραγωγή αυτή τα λάπια, η πάγκρασιους, τα φιλέτα, πώς τα λένε αυτά τα ψάρια στο Βιετνάμ. PCB, βαρέα μέταλλα και πάει λέγοντα, θα το ψάξετε αυτό και υπάρχουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την υγεία για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αν μπορούμε αυτό να το αποδείξουμε θα πούμε ότι δεν ε, πληρεί τις προϋποθέσεις και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μένει εκτός ενώσεως. Αυτά δεν μπορείτε να μου απαντήσετε συγκεκριμένα. der zwei η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι για να απαντήσει αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την τελευταία ερώτηση. Εγώ είμαι στι υπηρεσίε Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για τη θάλασσα και δεν μπορώ να σα απαντήσω από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσια Υγεία, ΣΑΝΚΟ για τις επιθεωρήσεις ε, προβλέπετε φέτος να ξεκινήσουν για τις προτεραιότητες και την ταξινόμησή τους. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Αν θέλετε θα διαβιβάσω αρμοδίως το ερώτημα. Σε ό,τι αφορά την υγεία των ζώων και την προστασία των καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε βεβαίως, είναι οι μόνες νομοθεσίες που μας επιτρέπουν σήμερα να επιβάλλουμε περιορισμούς στις ε, εμπορικές συναλλαγές για τα ζώα έχουμε μια νέα οδηγία για την ε, προστασία ε, των οργανισμών των υδρόβιων, ψάρια και οστρακοειδή στις υδατοκαλλιέργειες και έχουμε ένα ολόκληρο μηχανισμό πιστοποίησης για την παραγωγή και τις ε, ανταλλαγές που μπορούν να προωθήσουν κάποιες αρρώστιες. Αυτό υπάρχει, αλλά ισχύει μόνο για κάποιες ασθένειες που αναφέρονται σε ένα κατάλογο και ε, συνιστούν κίνδυνο ε, για τη δημόσια υγεία. Αυτά υπάρχουν. Ε, αλλά μιλάμε για κάποια είδη στην Ευρώπη, για κάποιες ασθένειες, δεν καλύπτουμε όλες τις ασθένειες, στα πλαίσια των παγκοσμίων συναλλαγών που καλύπτονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Ζώων. Θα έχετε ακούσει εδώ, είναι το Διεθνές Γραφείο Επιζωτιών, ε, που ασχολείται ακριβώς με την υγεία των ζώων, με την υγεία επαναλαμβάνω, όχι την ευημερία. Αμυγός με την υγεία. Το διεθνέ Γραφείο Επιζώτιων τώρα για την προστασία του καταναλωτού υπάρχει ένα σύστημα με δειγματοληψίες και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ε, επιθεωρήσεις, ε, πιστοποιήσεις και αντιστοιχίες σε τρίτες χώρες. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποια είναι τα προγράμματα των επιθεωρητών, δεν ξέρω αν φέτος θα πάνε στο Βιετνάμ ή όχι. Πάντως θα διαβάσω και αυτό το ερώτημα. Νομίζω όμως εδώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διακάκριση. Υπάρχει και μια εθελούσια πιστοποίηση έγινε λόγος για τις βιολογικές υδατοκαλλιέργειες, οι οργανικές τις λένε στα αγγλικά. Από πέρυσι υπάρχουν προδιαγραφές ευρωπαϊκές και είμαστε τώρα σε ένα σύστημα που είναι βασισμένο σε κάποια εθελούσια πρότυπα, όπως και για το υπόλοιπο. Και από εκεί και πέρα οι φορείς της αγοράς και εισαγωγή και οι ευρωπαίοι παραγωγοί μπορούν με ένα σύστημα ανεξάρτητης πιστοποίησης να αποδείξουν ότι τα κριτήρια γίνονται σεβαστά. Και τέλος, για το γενικό όρο αυτό της ε, πιστοποίησης, ε, ξέχασα να σας πω, στο ΦΑΟ γίνεται μια προσπάθεια για να ε, έχουμε παγκόσμιο ορισμό του τι εστί αηφόρους υδατοκαλλιέργεια. Στα μέσα Φεβρουαρίου επίκειται συνεδρίαση στο ΦΑΟ τεχνική εμπειρογνωμόνων για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αλλά βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα γίνει λόγος για ελάχιστα κριτήρια για παγκόσμια συνένεση. Και βεβαίως η κατάσταση και η οικονομική και η οικονομική και περιβαλλοντική διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, να προωθούμε τα δικά μας κριτήρια και τις τιμές και τις αξίες για την προστασία του περιβάλλοντος οπωσδήποτε. Και νομίζω, Πρόεδρε, ότι απάντησα σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγκήτρια. Ναι, πολύ σύντομα. Χαίρομαι πολύ που έγινε ευρύτατη συζήτηση και μίλησαν και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Θυμάστε ότι κάναμε και ολόκληρη συζήτηση αν έπρεπε να γνωμοδοτήσουμε, κάνει όχι. Νομίζω καλή ιδέα ήταν να κάνουμε γνωμοδότηση και ε, προσφέρθηκα κι εγώ εθελοντικά να γράψω ένα τέτοιο κείμενο. Λέτε ε, κάποιοι συνάδελφοι ότι είναι αρνητική η προσέγγιση μου. Το ξέρω ότι υπάρχουν και πολλά θετικά και θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε, αλλά σας είπα ότι είχα τόσο μεγάλο περιορισμό και είπα ότι τα θετικά θα τα πει η Επιτροπή Αλίας. Οπότε θεώρησα ότι ήταν καλό εγώ να αναφέρω τα προβλήματα από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής. Και αν είναι αυτό μια λύση και μια απάντηση στην υπεραλίευση, εντάξει, αλλά να τονίσουμε και τα αρνητικά. Νομίζω ότι ο κύριος Σαφ μίλησε για τα οικολογικά χαρακτηριστικά της ε, υδατοκαλλιέργειας. Καλή ιδέα. Πολλοί συνάδελφοι μίλησα για θέμη του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες και είπε κάτι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Και είναι αυτός ένας από τους λόγους που έχω βάλει το σημείο 4 στην έκθεσή μου, έτσι ώστε να ζητήσω άδεια κυκλοφορίας ε, για συγκεκριμένα προϊόντα. Γιατί, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει πρόταση του Κοινοβουλίου στον κανονισμό Novel Food για τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον και η ευημερία των ζώων. Ένα τμήμα το λύνει αυτό του προβλήματος. Αν οι συνάδελφοι έχουν καλύτερη ιδέα, τους παρακαλώ να απευθυνθούν σε μένα και να μου το πούν. Τι άλλο έχω εδώ. Α, μήπως θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο χώρο στη διάθεση του τα ψάρια, όπως είπαμε και για τα κοτόπουλα. Αυτό διαφέρει βέβαια από ε, είδο σε είδο του ψαριού. Δεν γνωρίζω τα δεδομένα και τα στοιχεία. Υπάρχουν, δεν τα έχω υπόψη μου. Θα χρειαστεί μεγαλύτερη μελέτη. Πολλέ ε, οργανώσει ευημερία των ζώων έχουν τέτοια στοιχεία. Και συμφωνώ και με την κυρία Λεπάζ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θεμελιώδη βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, καλό είναι να λύσουμε το θέμα της υπεραλίευσης, αλλά να μην το λύσουμε προκαλώντας πολύ περισσότερα και άλλα προβλήματα. Γιατί είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντος εμείς και ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ε, προσβλέπω στην εργασία σας και ελπίζω να μπορέσω να υποστηρίξω και να δεχτώ πολλές από τις ιδέες σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λιωτά. Κατεθουσιασμένη από τη μεγάλη απήχηση που είχε το θέμα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό. Έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες 22 2 Φεβρουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 23 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή. Και πάμε στα σημεία 5 και 6 τώρα. Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. Είναι το λεγόμενο πακέτο για τα φάρμακα, ένα τμήμα σε πρώτη ανάγνωση. Λίντα Μακάβεν, η και έχει το λόγο. Um, thank you, Chair. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όσους δεν βρίσκονταν εδώ την τελευταία φορά που συζητήσαμε, τον Νοέμβριο, να θυμίσω ότι αυτέ τι δύο εκθέσει θα τι εξετάσουμε μαζί για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Μιλάμε εδώ για ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για να παρακολουθούμε την ασφάλεια των ε, φαρμάκων εφόσον έχουν εξοδοτηθεί και εγκριθεί να διατεθούν στην αγορά. Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων ε, θα χάνουν τη ζωή του, οι ασθενούν λόγω της κακή χρήση φαρμάκων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της δημόσιας υγείας αυτό. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπήρξαν δίκες και καταδίκες και αποφάσεις για κάποια από τα φάρμακα και προέκυψε και ένα σύστημα κανόνων ε, το οποίο έχει να κάνει με τη χρήση των φαρμάκων, ε, το... Θα θυμάστε φάρμακα τα οποία τη δεκαετία του 60 μετά τη χρήση τους διαπιστώθηκε ποιες ήταν οι παραενέργειές τους και τι μέρη να χρειάστηκε να λάβουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Εδώ προτείνονται δύο επιλογέ. Το σύστημα τη αμοιβαία αναγνώριση και τη αποκεντρωμένη διαδικασία για τα κράτη-μέλη, όπου μια χώρα συντονίζει τα κράτη-μέλη και τη συνεισφορά του και μετά χρησιμοποιείται μια κεντρική διαδικασία για την περίπτωση όπου μια φαρμακοβιομηχανία καταθέτει την αιτησή της στον, ε, ναι, τον Ευρωπαϊκό Φαρμακευτικό Οργανισμό. Εδώ για νέα προϊόντα όπως ε, τα φάρμακα για τον ε, ιό του AIDS, ή φάρμακα που φροντίζουν για την μη επιδείνωση του νευρικού συστήματος, όλα αυτά είναι νέα φάρμακα που μπορούν να περάσουν από την κεντρική διαδικασία. Τα κριτήρια για την κεντρική διαδικασία ορίζονται ακριβώς στον κανονισμό. Η Επιτροπή προτείνει να, να ενημερωθούν οι κανόνες τόσο της οδηγίας όσο και του κανονισμού, αλλά τα στοιχεία που προσπαθεί εδώ να καλύψει είναι κοινά και στην οδηγία και στον κανονισμό. Έτσι λοιπόν τα σχόλιά μου αφορούν και τα δύο αυτά νομοθετήματα. για να έχουμε ένα καλό σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης είναι να παρακολουθούμε και να ενημερωνόμαστε για τις παρενέργειες. Μόλις δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να μπορούμε για το συγκεκριμένο φάρμακο να αλλάξουμε την αποτίμηση που υπάρχει για τις κινδύνους και τις απειλές που ενέχει. Να αλλάξουμε τη δοσολογία που προβλέπεται ή, στην περίπτωση σοβαρών παρενεργειών, να προτείνουμε την απόσυρσή του από την αγορά. Ολοσχερός. Έτσι λοιπόν το πώς καταγράφονται οι παρενέργειες αυτές, οι ADR όπως ονομάζονται, οι φαρμακευτικές παρενέργειες, ε, είναι σημαντικό. Μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις που το κοινό εντοπίζει ή οι επαγγελματίες του τομέα υγείας ή οι ίδιες φαρμακοβιομηχανίες. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αυτό ακριβώς αφορά το νομοθέτημα εδώ. Πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο εντοπίζει τις σοβαρές παρενέργειες και πώς αυτές θα παρακολουθούνται για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας. Το κεντρικό σύστημα λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια και κάποια κράτη-μέλη επίση έχουν συνεργαστεί εδώ και κάποια χρόνια και η Επιτροπή σημειώνει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τον τρόπο που συνεργαζόμαστε για τι παρενέργειε και τη σχετική νομοθεσία. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κοινό κτήμα τη γνώση που διαθέτουμε για τι παρενέργειε, τόσο καλύτερο. Δηλαδή το να εργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικό διότι κάποια παρενέργεια είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί εάν τι πληροφορίε που λαμβάνουμε από διαφορετικέ χώρε φροντίζουμε να τι συλλέγουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα τέτοιο κεντρικό σύστημα συγκέντρωση τη γνώση, μια βάση δεδομένων που ονομάζεται Eurovigilance. Eurovigilance, ε, η οποία συγκεντρώνει ε, στοιχεία για παρενέργειες και από τις εταιρείε και από τις δημόσιες αρχές στα κράτη-μέλη και εδώ, εάν δούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία του νομοθετήματος που μας απασχολεί, να υπογραμμίσω κάποιες από τις βασικές πτυχές. Συμφωνώ εδώ με αυτά που προτείνει επιδιώκει η Επιτροπή για αλλαγέ, Πρώτα απ' όλα, συνολικά, το ζήτημα της ε, δομής των επιτροπών. Επιτροπών που είναι υπεύθυνε για το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης. Εδώ υπάρχει μια Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης που είναι όμως αρκετά αδύναμη προς στιγμή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί, λέει η Επιτροπή, η Επιτροπή αυτή και να δημιουργηθεί και μια ειδική επιστημονική επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φαρμακευτικού Οργανισμού. Η Επιτροπή προτείνει να υπάρξουν επιστήμονε από τα βασικά κράτη-μέλη που να αντιπροσωπεύουν τα κράτη-μέλη για να επιδιώκουν κοινού στόχου Ακούγοντα τώρα την αντίδραση των κρατών μελών, πιστεύω ότι ναι, πρέπει να υπάρχει μια ε, ε, επιτροπή που να αντιπροσωπεύει του πάντε σε επίπεδο ΕΜΕΑ, διότι ακριβώ υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε στο κοινό για τα ζητήματα δημόσια υγεία. Είναι λοιπόν προφανέ ότι κάθε χώρα θα θέλει να συμμετέχει σε μια τέτοια επιστημονική επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να προσθεθεί σε αυτό και η παρουσία δικαστικών εκπροσώπων από την ομάδα ασθενών και από την ομάδα επαγγελματιών του τομέα υγείας. Και αυτό σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες επιτροπές του ΕΝΕΑ. Εάν δεχτούμε λοιπόν η επιτροπή αυτή να γίνει πιο αντιπροσωπευτική για όλα τα κρατημέλη, η Επιστημονική Επιτροπή, τότε θα μπορούσαν να αλλάξουν και αρμοδίτητέ τη. Ο τρόπο που έχει θεωρήσει το θέμα αυτό η Επιτροπή είναι να συγκεντρώνει στοιχεία η Επιτροπή αυτή και να τα παραπέμπει στην ανώτερη από αυτήν την επιτροπή και μετά να ακολουθεί την τυπική διαδικασία. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι ότι αν έχουμε ένα αντιπρόσωπο αναγκαίο μέλο, να μπορεί ο ίδιο ο αντιπρόσωπο να εκφέρει συστάσει για τι παρενέργειε και το τι παρακολούθηση θα πρέπει να δοθεί στο θέμα ώστε η εξουσιοδότηση των φαρμάκων και η παρακολούθηση του πώ αυτά ενεργούν στου ασθενεί, να είναι κάτι που θα γίνεται από κοινού. Οι αποφάσεις λοιπόν τη ε, Επιτροπή αυτή τη ΠΡΑΚ να γίνεται κατεξοχήν εκεί και οι υπόλοιπε επιτροπέ, αν θέλουν να μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση απόφαση. Τώρα, τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Οι κυβερνήσει με τα χρόνια έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά δικά του μεμονωμένα συστήματα φαρμακοταγρύπνηση και πολλέ φορέ αμελούν στη συγκέντρωση των πληροφοριών και στην ε, διοχέτευσή τη προ μια κοινή τράπεζα ευρωπαϊκή. Εδώ, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πολύ γρήγορα να μπορούμε να εντοπίσουμε τις παρενέργειες από τη μια χώρα στην άλλη. Θα πρέπει δηλαδή τα κάτι μέλη να μπορούν να ενημερώσουν για το τι συμβαίνει στη χώρα τους, αλλά και να παραδεχτούν την ανάγκη συγκέντρωσης των δεδομένων σε εκείνη βάση. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται ένα συμβιβασμό μεταξύ του αυτού που προτείνει τώρα η Επιτροπή. Δηλαδή, εάν μια εταιρεία έχει εντοπίσει παρενέργεια ή ενημερωθεί για παρενέργεια, να ενημερώνει τότε την, επιστημονική, την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων, εγώ θα έλεγα αμέσω η τράπεζα να ενημερώνει με τη σειρά τη ε, τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν και αυτά να παρακολουθούν εάν θα υπάρξει και στην περίπτωσή του παρενέργεια. Το συζητήσαμε διαμακρών με το Συμβούλιο για την φαρμακοπαγρύπνηση. Ε, η Επιτροπή εδώ αυτό που προτείνει είναι όπως τώρα μόνο σοβαρές παρενέργειες να, να επισημένονται στο κεντρικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Δεδομένων. Η Επιτροπή λοιπόν προτείνει πλέον να αλλάξει αυτό και να, να εντοπίζονται τόσο σοβαρές όσο και λιγότερο σοβαρές παρενέργειες. Να φορτώνονται όλα τα στοιχεία στο κεντρικό σύστημα δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και με το Συμβούλιο. Και ακριβώς έτσι προχωρούν οι συζητήσεις μας το τρίτο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι οι εκθέσει για του ασθενεί. Εδώ υπάρχουν αρκετέ αμφισβητήσει γιατί η Επιτροπή προτείνει οι ασθενείς να μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι τα στοιχεία τους στην αρμόδια αρχή τους, εφόσον το θέλουν, και όχι στην ε, βάση δεδομένων της φαρμακοπαγρύπνησης. Αυτό προκαλεί κάποια σύγχυση, γιατί είχε προταθεί οι ασθενείς να μπορούν να πάνε απευθεία στην τράπεζα φαρμακοπαγρύπνησης. Αλλά τώρα προτείνεται η επαφή τους με την δημόσια αρχή, εφόσον υπάρχει σοβαρή παρενέργεια. Αυτό ήδη συμβαίνει σε πολλές χώρες. Στη δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ και καιρό δηλαδή από τη δεκαετία του 60, έπειτα στη Δανία και τις κάτω χώρες, από δεκαετία του 90, καθώς και στη Σουηδία και τη Γαλλία. Υπάρχει σύστημα για την ενημέρωση των ενώσεων ασθενών, οι οποίοι μετά φροντίζουν να παραπέμπουν τα στοιχεία στην αρμόδια δημόσια αρχή. Μετά την έρευνα που έκανα και από όσα γνωρίζουν και οι σκιώδεις εισηγητές για αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την Επιτροπή στην ε, υποβολή από τους ασθενείς, αλλά όχι μόνο μέσω μηχανισμού του διαδικτύου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα αυτό και θα πρέπει να γίνει εύκολη υποβολή στοιχείων από τους ασθενείς. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό φυλάδιο που να διατίθεται στους ασθενείς και η αρμόδια αρχή να το λαμβάνει άμεσα και εύκολα να το, ε, και γρήγορα να το διεκπαιρεώνει να εξετάζει τα στοιχεία. Ένα άλλο τομέα που έχει προκαλέσει πολλέ αμφισβητήσει είναι η πρόταση τη Επιτροπή για τα εντατικώ ε, παγκόσμια προϊόντα. Εδώ μιλάμε για φάρμακα που έχουν διατεθεί στην αγορά πρώτη φορά, για πρώτη φορά ίσω και οι εταιρείε πρέπει να κάνουν μελέτε παρακολούθηση. Η περίοδος εντατικής επαγρύπνησης λοιπόν για την περίπτωση παρουσίασης παρενεργειών σημαίνει ότι παρόλα αυτά τα φάρμακα λαμβάνονται από ασθενεί. Η Επιτροπή λοιπόν προτείνει να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου να ενημερώνονται οι ασθενεί για τη λήψη τέτοιων προϊόντων. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζεται στο σχετικό φυλάδιο ενημέρωση των ασθενών κατά την άποψή μα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι φοβούνται ότι αυτό θα δημιουργήσει άγχο και ε, αναστάτωση στους ασθενείς. Αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι ασθενείς πρέπει να είναι ενήμεροι. Εγώ από τις φαρμακοβιομηχανίες με τις οποίες συζήτησα γνωρίζω ότι δεν είναι ικανοποιημένε με τέτοια πρόταση. Και το επιχείρημά τους είναι ότι αν οι ασθενείς δουν κάποιο σύμβολο που λέει ότι το φάρμακο αυτό παρακολουθείται εντατικώς, μπορεί να φοβηθούν και να μην πάρουν τελικά το φάρμακο. Όμως όλα τα φάρμακα μπορεί να έχουν ωφέλειες ή όχι όταν τα λαμβάνει κανεί. Κανένα φάρμακο δεν είναι 100% ασφαλέ. Κάποιο μπορεί να παρουσιάσει παρενέργεια σε ένα φάρμακο, κάποιο άλλο δεν θα παρουσιάσει. Οπότε, κατά την άποψή μου, πρέπει να στηρίξουμε την Επιτροπή στην πρότασή τη. Και να ενημερώνουμε παρόλα αυτά του ασθενεί ότι λαμβάνουν φάρμακο εντατικώ παρακολουθούμενο. Τώρα, αν θα πρέπει να το ονομάσουμε το φάρμακο αυτό εντατικώ επαγρυπνούμενο, δεν είμαι βέβαιη. σω απλώ να λέμε ότι πρόκειται για ένα νέο προϊόν. όμω. Νομίζω ο τρόπος που θα ενημερώνουμε τον ασθενή για το γεγονό ότι λαμβάνει τέτοιου είδους προϊόν είναι χρησιμοποιώντα ένα μαύρο τρίγωνο, ανάποδο μάλιστα. Αυτό το τρίγωνο ήδη χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και μάλιστα υπάρχει στο φυλάδιο ενημέρωση των επαγγελματιών του τομέα υγεία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στο φυλάδιο των ασθενών. Ένα άλλο τομέα που προκαλεί αμφισβητήσει, το συζητήσαμε με πολλού από του φορεί, είναι οι βασικέ πληροφορίε ασφάλεια. Η Επιτροπή λέει ότι όταν οι ασθενεί λάβουν το φυλάδι ενημέρωση των ασθενών, περιέχει υπερβολικά πολλά δεδομένα. Η πρόταση είναι λοιπόν τα βασικότερα, τα σημαντικότερα, να χρησιμοποιούνται σε, να συμπεριλαμβάνονται σε ένα μαύρο πλαίσιο ή με έντονου χαρακτήρε. Οι ομάδε όμω ασθενών, οι ενό ασθενών, οι γιατροί, οι επαγγελματίε τη υγεία έχουν ανάμεικτε απόψει. Λένε ότι αυτό που μπορεί να είναι σημαντικό για τον ένα ασθενή μπορεί να μην είναι για τον άλλο. Πώ θα κάνουμε εμεί τη διάκριση, πώ θα επιλέξουμε τα σημαντικά δεδομένα εμεί για το κάθε προϊόν. Και κάποιοι άλλοι επίση υποστηρίζουν ότι τα ίδια τα φάρμακα στι οδηγίε χρήση περιέχουν τόσε πολλέ οδηγίε τελικά που αν τι διάβαζε κανεί όλε δεν θα το παίρνει ποτέ το φάρμακο. Οι εταιρείε προσφέρουν όση γνώση μπορούν για το κάθε φάρμακο για να είναι καλυμμένε, αλλά τελικά οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι όσο περισσότερο διαβάσει κανεί τα σχετικά φυλάδια, τόσο πιο σοφό γίνεται και η ουσία είναι να πάρει και το φάρμακο. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του χαπιού εδώ σε αυτή την οδηγία. Πάντω, η δική μου εντύπωση είναι ότι ο Ευρωπαϊκό Φαρμακευτικό Οργανισμό το μήνα αυτό που ξεκίνησε και ήδη είχε αρχίσει πριν από τα Χριστούγεννα, οργάνωσε διαβουλεύσεις ε, για να δει πώ θα διαμορφωθεί ακριβώ το φυλάδιο ενημέρωση των ασθενών. Στι προτάσει λοιπόν που κάνω προ την Επιτροπή φροντίζω αυτό να ληφθεί υπόψη και αναμένουμε διακαώς το φυλάδιο ενημέρωση των ασθενών καθώ και τι απόψει των συναδέλφων ώστε να βεβαιωθούμε ότι ένα τέτοιο φυλάδιο θα είναι πραγματικά ενημερωτικό και να μην απαριθμεί απλώς όσα μπορεί πιθανώς να συμβούν σε, κάποιοι, σε κάποιον. Κάτι άλλο από τις βασικές προτάσεις της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ένα εθνική, δημιουργία εθνικών ιστοτόπων. Αυτό γίνεται σε επίπεδο Επιτροπής ΠΡΑΚ, ώστε να μπορούν οι ασθενείς να παρακολουθούν τις συζητήσει βάσει των δεδομένων που συλλέγονται στην Τράπεζα Δεδομένων. Αλλά τα δεδομένα αυτά λέγεται ότι θα πρέπει να διατίθενται και στο κοινό. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον κάποια δεδομένα μπορούν να δημοσιοποιούνται ή όχι. Στι Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που δημοσιεύονται, δημοσιοποιούνται στην, παρά στην Ευρώπη και εδώ καλωσορίζουμε τι σχετικέ προτάσει τη επίτροπή, αλλά υπάρχουν και εμπορικώ μάλλον εμπιστευτικέ πληροφορίε, καθώ και αυτέ που μπορεί να μην ευσταθεί να δημοσιοποιηθούν. Βάσει λοιπόν των ε, προτάσεων της Επιτροπής στηρίζω την ε, διενέργεια δημόσιων ακροάσεων για τη χρήση νέων φαρμάκων, πράγμα που γίνεται και σε πολλές άλλες χώρες καθώς και στις ΗΠΑ. Και κάτι άλλο που μου εντόπισαν συνάδελφοι είναι πώς θα χρηματοδοτήσουμε την φαρμακοπαγρύπνηση και πώς θα φροντίσουμε να λειτουργήσει. Σε κάποιες χώρες το σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης, οι επιτροπές τους, οι εθνικές δημόσιε αρχές ε, χρηματοδοτούνται από τα ε, δημόσια κονδύλια, τα κρατικά κονδύλια. Διότι αν ζητήσει κανείς από τις φαρμακοβιομηχανίες να καταβάλουν ε, τη χρηματοδότηση αυτή προς τη δημόσια αρχή και κατά συνέπεια προς το σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης, τελικά οι πληροφορίες θα είναι αντικειμενικές. Στη χώρα μου δεν ισχύει αυτό. Το σύστημα της φαρμακοπαγρύπνησης χρηματοδοτείται μέσω φορολόγησης των φαρμακοβιομηχανιών. Ε, σε ένα πρόσφατο νομοθέτημα φροντίσαμε να χωρίσουμε τη χρηματοδότηση του ΕΜΕΑ. Να υπάρχει χρηματοδότηση εν μέρει από το προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπόλοιπο μέρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να χρηματοδοτείται από φόρο των φαρμακοβιομηχανιών. Ε, στοιχεία έγκριση, καταγραφή και ούτω καθεξή. Όμω εδώ πρόκειται ένα ψευδή διαχωρισμό του προπολογισμού. Γιατί το ΕΜΕΑ τελικά είναι ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Εάν κοιτάξει κανεί τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, α πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία, υπάρχει ένας δασμός, ένας φόρος που αξιοποιείται για την χρηματοδότηση της φαρμακοαπαγρύπνησης και δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία των επιτροπών φαρμακοαπαγρύπνησης. Νομίζουμε ότι την ανεξαρτησία αυτή μπορούμε να την εξασφαλίσουμε και με άλλους τρόπους. Δεν είναι μόνο η ε, χρηματοδότηση το κριτήριο που θα καθορίσει το πώς θα δουλέψουν. Εδώ λοιπόν πραγματικά στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλά ακόμη ζητήματα, λεπτομέρειες ενδεχομένως, τις οποίες ίσως να μην θίξω προς στιγμήν, αλλά σε κάποια άλλη ευκαιρία. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που ήθελα να συζητήσω με τους συναδέλφους και αναμένω τα σχόλιά τους. Äh, Σας ευχαριστώ. Σημαντικό θέμα. Μεγάλης προτεραιότητας. Στην ε, ατζέντα της ε, πολιτικής υγείας, τα ασφαλή φάρμακα δηλαδή. Υπάρχει μια αγορά των 27 χωρών μελών που υποτίθεται ότι θα συνεργαστούν και συνεργάζονται για την παραγωγή των φαρμάκων. Ακούσαμε που βρίσκονται τα σημεία τριβής και τα ελλείμματα. και όπου συμβάντα σε μια χώρα μέλος πρέπει να καθίστανται γνωστά αμέσως σε όλες τις άλλες χώρες μέλη. Ζητούν το λόγο τώρα οι σκιώδεις και πρώτη κυρία Πιλάρα Γιούσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ και την εισηγήτρια την κυρία Μακάβαν που πράγματι έθεσε επιτάπητος τα ε, επίμαχα σημεία που κρύβονται σε αυτή την νομοθεσία. Σε τελική ανάλυση αποσκοπεί στη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα για ένα σύστημα προς όφελος όλων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε γενικές γραμμές είναι και καλή και ε, αποδεκτή. Η κυρία Μακάβαν ακριβώς ε, ανέφερε τα πιο επίμαχα σημεία όπως σας είπα και σε ό,τι αφορά το πρώτο άρθρο και της οδηγίας και του κανονισμού, εγώ δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα με την εισηγήτρια. Θα πρέπει η Συμβουλευτική Επιτροπή να έχει τις σωστές αρμοδιότητες για να ε, εκτιμήσει τον κίνδυνο στην φαρμακοεπαγρύπνηση, γιατί επιφορτίζεται με αυτό το έργο. Συμφωνώ επίσης να εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη, οι ασθενείς και ε, το υγειονομικό προσωπικό στο σχέδιο έκθεσης της η συγγήτρια επιθυμεί η Επιτροπή αυτή να μην είναι συμβουλευτική, αλλά να κάνει και συστάσεις. Και μιλάει για την Επιτροπή ε, για τα ανθρώπινα φάρμακα που μπορεί να απορρίψει μόνο μία σύσταση μόνο εφόσον αυτό στοιχειοθετείται από επιστημονική ιατρική γνώση σε σχέση με τη δημόσια υγεία. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε περίπτωση που αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν δέχεται τις προτάσεις της άλλης Επιτροπής για τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, ποιος έχει τον τελευταίο λόγο. Αν διαφωνήσουν αυτές οι δύο επιτροπές, γιατί και τα επιστημονικά στοιχεία ε, χωρούν αμφισβήτηση. Αυτό θα ήθελα ε, να μου πείτε ποιος θα έχει το καθοριστικό λόγο για να αποφασίσει ποιος έχει δίκιο. Είναι η μόνη επιφύλαξη και αμφιβολία που έχω. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ απολύτως. Και για τη βάση δεδομένων, επίσης συμφωνώ με την κυρία Μακάβων, θα πρέπει να υπάρχει εγγυημένη ταυτόχρονη πρόσβαση από την αρμόδια αρχή ε, του κράτους μέλους, όπου ε, είδαμε την παρενέργεια, και να συντονίζονται οι βάσεις δεδομένων και όλες οι δράσεις στη συνέχεια. Επίσης θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα τεχνικά και τα ανθρώπινα μέσα και οι πόροι που θα διατεθούν για να υλοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Πολύ ωραία τα βλέπουμε στα χαρτιά, αλλά στην πράξη τι θα γίνει. Και αν προβλέπονται μεταβατικοί κανόνες για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, μπορεί αυτό να το υπονομεύσει και την αποτελεσματικότητά του και ταυτόχρονα είπαμε θα πρέπει να διαβάζονται οι παρενέργειες, να ενημερώνονται όλοι και η ενημέρωση των ασθενών τώρα γίνεται από τις αρμόδιες αρχές ή από τη βάση δεδομένων. Εντάξει, συμφωνώ και σε αυτό απολύτως. Θα πρέπει να υπάρξει ένα μικρό φίλτρο γιατί όλοι οι ασθενείς δεν έχουν την ίδια γνώση, ούτε ίση είναι μεταξύ του, ούτε, ούτε μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιοι τον εαυτό του ω άρρωστο με τον ίδιο τρόπο και η πληροφόρηση μπορεί να του οδηγεί ενδεχομένω σε σύγχυση, να μην τους προσφέρει τίποτα καινούριο όταν είναι αντιφατική. Και για τη διεκτυακή πύλη που πρότεινε η συγγήτρια συμφωνώ επίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να ε, βάλει νέα πληροφορία, ε, λέει μια σύνοψη των βασικών πληροφοριών, μια περίληψη για τη χρήση του φαρμάκου, ε, θα πρέπει να πούμε ότι και το 2003 όταν θεωρήθηκε η φαρμακευτική νομοθεσία συζητήθηκε το θέμα αυτό και καταλήξαμε στο ότι το ενημερωτικό φυλάδιο θα πρέπει να έχει τις σημαντικές θεμελιώδεις ε, πληροφορίες και ευανάγνωστες. Τώρα βάλουμε την περίληψη της περίληψης έχει περισσότερα μειονεκτήματα από πλεονεκτήματα. Θα είναι και υπερβολικός φόρτος και για τα εργαστήρια και για τους οργανισμούς φαρμάκων. Και στη συνέχεια μπορεί να είναι αναποτελεσματικό να διαβάσουν μόνο την περίληψη οι ασθενείς και όχι ολόκληρο το φυλάδιο, αυτό είναι αντιπαραγωγικό, γιατί θα διαβάσουν μόνο τα αρνητικά, το πιο αρνητικό. Μα όλα τα φάρμακα έχουν και θετικά, έχουν και αρνητικά ενδεχομένω ανεπιθύμητε ενέργειε και παρενέργειε και αν δεν δείξει και τρίτον, η, ουσιαστική, η βασική προφόρηση μπορεί να διαφέρει από τον ασθενή σε ασθενή, ανάλογα με την ηλικία του, τη μόρφωσή του, την ενημέρωσή του, την κατάστασή του. Και τελικά κινδυνεύουμε να τον ε, κατακλείσουμε τον ασθενή με άχρηστες προφορίες. Ε, λοιπόν, σας ανέφερα. Τα φυλάδια έτσι και ε, είναι δύσκολα να τα καταλαβούν οι ε, καταναλωτέ, τι οδηγίε που είναι μαζί με το φάρμακο και δεν θέλουμε να του οδηγήσουμε σε μεγαλύτερη σύγχυση. Και μια λύση θα μπορούσε να να κάνει η μελέτη για ε, το ενημερωτικό αυτό ε, φυλάδιο σημείωμα που συνοδεύει το φάρμακο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνει πρόταση. Η συγκήτρια μίλησε για ένα δεστραμμένο μαύρο τρίγωνο Απλό είναι αυτό, εύκολο να το καταλάβει όλος ο κόσμος ότι το φάρμακο αυτό είναι που παρακολούθηση και καλή ιδέα τη βρίσκω. Και ένα τελευταίο, για τις δημόσιες ακροάσεις, οι συνεδριάσεις. Υπάρχει πάντα ε, το διώνυμο κόστος-οφέλεια όταν μιλάμε για τέτοιες δημόσιες ακροάσεις. θα πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος της Επιτροπής για τα φάρμακα, για ανθρώπινη χρήση, του οργανισμού φαρμάκου, για να μην μιλάμε μόνο για τους κινδύνους, αλλά και για το όφελος. Γιατί πολύ συχνά ο ασθενής, όταν τονίζουμε τόσο πολύ τα αρνητικά ενός φαρμάκου που είναι καλό για την υγεία του, ε, δεν θα το πάρει και θα βλάψει την υγεία του. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την εισηγήτρια και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παρά. Dankeschön. Antonia Paravadova. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to congratulate the rapporteur. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να συγχαρώ την εισηγητρία την κυρία Μακέβαν για τη δουλειά της. Σίγουρα ένα όριμο σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης χρειάζεται την καλύτερη δυνατή ποιότητα και τις αυστηρότερες δυνατές προδιαγραφές. Συμφωνούμε λοιπόν με τις περισσότερες από τις προτάσεις της, όμως το σχέδιο της έκθεσής της μπορεί περαιτέρω να συμπληρωθεί με κάποια στοιχεία για τα βασικά σημεία σχόλια του κανονισμού και της οδηγίας, ιδίως για τις βασικές αρχές διαφάνεια, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Νομίζω το στοιχείο τη εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικό για όλους του εμπλεκόμενου φορεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο ασθενής προφανώς πρέπει να μπορεί να εμπιστευτεί την αγωγή που του χορηγείται. Οπότε δεν ανάγκη να θυμίζουμε όταν μιλάμε για φάρμακα, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ποιο είναι ο κίνδυνο και ποια είναι η ωφέλεια για του ανθρώπου και του πολίτε από άποψη συμπεριφοράς και μόνο, δεν πρέπει να αποθαρρύνουμε τους ασθενείς να διακόπτουν την αγωγή τους ή να πάβουν να απόσχουν από μια αγωγή λόγω κακής διατύπωση ή κακής ενημέρωσή τους. Οι δημόσιες, οι εθνικές αρχές λοιπόν και η βιομηχανία θα πρέπει να στηρίξουν το νομοθέτημα αυτό και να συμμετάσχουν πλήρως τα όσα αυτό προβλέπει. Έχω κάνει συγκεκριμένε προτάσει και συστάσει και τι έχω οργανώσει σε τρει βασικέ ομάδε. Πρώτα απ' όλα για την Επιτροπή Αποτίμηση του Συστήματο Φαρμακοεπαγρύπνηση. Νομίζω η πρόταση πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Απλώ νομίζω ότι 27 εκπρόσωποι κρατών μελών συν τρεις ε, εκπρόσωποι από τις ενώσεις ασθενών και από το τομέα υγείας ίσως κάνει πολύ ευρεία την ομάδα. Εφόσον υπάρχουν διαρκείς διαφωνίε μεταξύ των δύο επιτροπών επίσης του ΕΜΕΑ, ποιο θα είναι τελικά υπεύθυνο για την τελική απόφαση και ποιε θα είναι οι συνέπειε μια διαφωνίας για τον, τέτοιες διαφωνίες για τους ασθενείς, τη δημόσια γνώμη και τη διαδικασία επίλυση των διαφορών θα προβλεφθεί. Επίση, οι δημόσιε ακροάσει είναι σημαντικό στοιχείο για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη και η συνολική διαφάνεια για το σύστημα φαρμακοπαθρύπνηση. Όμω, αν δει κανεί ε, τι τέτοιε ακροάσει έχουν ε, οργανωθεί από του ε, φαρμακευτικού οργανισμού ω τώρα, θα καταλάβουμε ότι Τέτοιε ακροάσει είναι απαραίτητε. Θα πρέπει λοιπόν τα μέλη τη CHNP και τη ΠΡΑΚ να συγκεντρώνονται και να οργανώνουν από κοινού τέτοιε ακροάσει. Και για να ωφεληθεί ακόμη περισσότερο το κοινό. Είναι σημαντικό για τέτοιου σκοπού να διασφαλίσουμε την συνεργασία του. Επίση, τα μέτρα που θα επηρεάσουν το φυλάδιο ενημέρωση των ασθενών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μια περίληψη των βασικών πληροφοριών και όπω είπε και η κυρία Αγιούζο, ήδη υπάρχει περίληψη και η Επιτροπή είπε ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ήδη ποιε πληροφορίε θα συμπεριλαμβάνει αυτή η βασική περίληψη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη ότι οι πληροφορίε που θα περιλαμβάνει το φυλάδιο ενημέρωση ασθενών είναι πληροφορίε που ούτω ή άλλω διέπονται από του κανόνε άλλη οδηγία. Είναι περίεργο όρο ούτω ή άλλω essential information, βασικέ πληροφορίε δεν ξέρουμε αν και ο ασθενή θα εκτιμήσει το γεγονό ότι οι υπόλοιπε πληροφορίε θα παρουσιάζονται ω απουσιώδει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δει με προσοχή η Επιτροπή. Επίση για τα εντατικώ ε, παρακολουθούμενα προϊόντα. Θα πρέπει οι ασθενεί να ενημερώνονται για το τι είδου φάρμακα παίρνουν, να ξέρουν αν αποτελούν αυτά αντικείμενο διαρκού και εντατική επαγρύπνηση, αλλά να μην προκαταλαμβάνονται. Να μην πιστέψουν ότι άλλα προϊόντα μπορεί και αυτά να μην παρακολουθούνται στον ίδιο βαθμό. Εδώ λοιπόν <clears throat> μια πρόταση που περιμένουν να βελτιώσουν οι φυσικοί ομιλητέ τη Αγγλική. Ίσως να πρέπει να χρησιμοποιήσουν έναν όρο όπω την μετά την εξουσιοδότηση παρακολούθηση. Post authorization monitoring. Τη διατύπωση βεβαίω θα τη δουν καλύτερα οι πλέον ειδικοί. Αν συμπεριλάβουμε μια τέτοια ιδέα, θα φροντίσουμε να βελτιωθεί και ο όρο που θα χρησιμοποιηθεί. Πάντω για τις νέες πληροφορίες και τη συμπερίληψή τους καθώς και τις νέες παρενέργειες που θα παρατηρώνται και θα εντοπίζονται με έντονους χαρακτήρες, αυτό μπορεί να προκαταλάβει πάλι τους ασθενείς. Να νομίζει ο ασθενής δηλαδή ότι η πληροφορία που φέρεται πιο έντονα είναι πιο σημαντική και εδώ δεν πρέπει να αποκλείσουμε βεβαίως ε, το να ανατρέξουμε σε μελέτες ε, της ε, βιωσόματος του φαρμάκου μετά την εξουσιοδότηση και την παρακολούθησή του σχετικά, καθώς και τα νέα επιστημονικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν εντωμεταξύ. Υπάρχουν εντατικές διαβουλεύσεις σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό και καλωσορίζουμε την ιδέα της έκθεσης να ενισχύσει μέσω της Επιτροπής το φυλάδιο ενημέρωση των ασθενών. Το πόσο μακριά θα πάμε όμω με αυτόν τον κανονισμό, με τα παραποιημένα φάρμακα και τη σχετική πρόταση, δείχνει ότι απαιτείται να έχουμε συνεπή προσέγγιση. Και η Επιτροπή να φροντίσει να καταλήξει σε συνεπή μεταξύ του συνεκτικά νομοθετήματα. Εδώ πρέπει να στηρίξω τη συνολική προσέγγιση της εισηγήτριας και για το σύστημα ε, υποβολή στοιχείων για τι παρενέργειε. Θα πρέπει οι ασθενεί άμεσα να μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία των παρενεργειών και οι βιομηχανίε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την τράπεζα δεδομένων. Και οι σχετικέ εκθέσει να ενημερώνονται διαρκώ. Τα έγγραφα να δημοσιοποιούνται. Μερικέ από τι εκθέσει αυτέ, τα στοιχεία δηλαδή που συλλέγονται, είναι πολύ σημαντικέ για του ασθενεί. Όμω, κάποιε μπορεί να αποτελούνται και από περισσότερε από χίλια σελίδε. Είναι άκρως τεχνικές πληροφορίε που περιλαμβάνονται στις έκθεσες αυτές. Μπορεί να αναφέρονται παρενέργειες ή άλλες, ε, άλλα στοιχεία που να μην σχετίζονται με το συγκεκριμένο φάρμακο που ο ασθενής καλείται να μελετήσει να ερευνήσει. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το προσέξουμε. Για την ενημέρωση για τις παρενέργειες και το του υπεύθυνε για την εξουσιοδότηση δημόσιε αρχέ, αυτές πιστεύω αμέσως θα πρέπει να ενημερώνονται και να, τις, ε, να τους δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, ώστε να έχουν και την ευκαιρία να αντιδράσουν άμεσα. Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις και τις συστάσεις που εγώ θα είχα να κάνω. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Marina ε, Ist irgendwie nicht da. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έρχεται σε ένα πολύ ε, επίκαιρο χρόνο και θα ήθελα να συγχαρώ και τη Λίντα Μακάβαν για τις προτάσεις που έκανε για ε, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι, λέω, πάρα πολύ επίκαιρο το κείμενο, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε ο κανονισμός και η οδηγία να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των ασθενών στα φάρμακα. Και όχι μόνο στα φάρμακα και το ε, σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης. Ε, νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα σημαντικό στάδιο, που είναι οι άδειε κυκλοφορίας. Θα πρέπει πραγματικά να ενισχυθούν οι κλινικές δοκιμές εκ των προτέρων. Δηλαδή, όταν παράγουμε ένα φάρμακο επιγόντως, γιατί είναι κερδοφόρο, αυτό θα πρέπει να είναι εξαίρεση. Το είδαμε πρόσφατα με τα εμβόλια της γρήψης. Και στην Ευρώπη, τελείως τυχαία, πολλοί κόσμος εμφανίζει επιφυλάξεις για τα εμβόλια και με τον τρόπο που κυκλοφόρησαν στην αγορά. Δηλαδή υπάρχει εδώ ένα ζήτημα ε, ως προς την εμπιστοσύνη και το, ε, κατά πόσο είναι αυλαβές ένα φάρμακο. Όχι, κάθε φάρμακο μπορεί να έχει παρενέργειες, δεν έχει απόλυτη ασφάλεια κανένα φάρμακο. Λοιπόν, για την άδεια κυκλοφορία. Πολύ σημαντικό ένα ε, σχέδιο διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να είναι η απόλυτη εξαίρεση. Μετά χρειάζεται καλή επιμελητεία και οργάνωση. Και επαναρχόμαστε στου εθνικού οργανισμού φαρμάκων. Πώ μπορούμε να φροντίσουμε έτσι ώστε οι παρενέργειε να δηλώνονται γρήγορα στις εθνικές αρχές και μετά στη ε, ε, ε επαγρύπνηση, στην βάσει δεδομένων είδατε τι έγινε με τη γρήπη είτε έναν ή ένα από χώρα σε χώρα. Άλλοτε δούλεψε καλά το σύστημα και οι γιατροί δήλωναν σωστά ε, τα κρούσματα και σε άλλες χώρες καθόλου. Δηλαδή θα πρέπει να ενισχυθούν οι κρατικές αρχές για να μπορούν οι γιατροί ε, ε, να δηλώνουν σωστά τις παρενέργειες, τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Στη Γαλλία ήμασταν στις 3.000 περίπου ε, παρενέργειες από 5 εκατομμύρια ε, άτομα που εμβολιάστηκαν. Σε άλλες χώρες είναι καμιά εκατοστή. Εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά ε, Άγγλοι, Γάλλοι, Ισπανοί έχουμε περίπου τις ίδιες παρενέργειες. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις κρατικές αρχές, χρηματοδότηση. Η Λίντα λέει ε, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ένα ιδιαίτερο τέλος ή από που το κρατικό προπολογισμό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάντως θα πρέπει κάπου να χρηματοδοτεί το δημόσιο για να ε, ενέχεται το κράτος σε αυτή την προσπάθεια ε, που γίνεται σε μια χώρα. Τώρα αυτό αν είναι τέλος, αν είναι φόρος, αν πληρώνεται ε, με τα φάρμακα, δεν ξέρω γιατί όχι. Αλλά προσοχή, στα διοικητικά συμβούλια της φαρμακοβιομηχανίας ε, ε, μάλλον σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια και τις διάφορες επιτροπές να μην κυριαρχεί σε αριθμό η φαρμακοβιομηχανία. Να υπάρχουν και εμπειρογνώμονες και γιατροί και ασθενείς, να μην κυριαρχούν οι εταιρείε. Τώρα, ε, η πρόσβαση στην ενημέρωση. Είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στην ενημέρωση και για το τι γίνεται στα εργαστήρια. Γιατί εκεί υποτίθεται ότι έχουμε το εμπορικό απόρριτο και οι εκθέσεις ε, εκτίμησης, αξιολόγησης ή κλινικές δοκιμές και παρενέργειες δεν δημοσιοποιούνται. Ενώ συχνά αυτό είναι δείκτες μελλοντικών παρενεργειών. Γι' αυτό έχει σημασία να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες και τα εργαστήρια και οι εθνικοί οργανισμοί. Και για το έντρα βιζιλάνς, όταν λένε ότι θα πρέπει να είναι δημόσιες αρχές ή ε, ειδικοί εμπειρογνώμονες, όχι, να, να ανοίξουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα πάει ένας ασθενής μόνος του. Εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών θα πρέπει να έχουν τη πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Και θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή να είναι αρκετή τα ευρεία αυτή η βάση δεδομένων για τη δήλωση, για την κοινοποίηση. Γιατί πολλές φορές όταν είναι κωδικοποιημένα δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά στοιχεία. Για τα φάρμακα συμφωνώ πολύ με τις προτάσεις που έγιναν, δηλαδή όταν κυκλοφορεί ένα νέο φάρμακο να μπαίνει ένα τέτοιο τρίγωνάκι ότι κοιτάξτε είναι ένα νέο φάρμακο, έχει περισσότερα ωφέλη από ρίσκα αλλά μάθετε ότι είναι νέο φάρμακο και χρειάζεται διαφορετική διαχείριση κινδύνου. Να γνωρίζει ο ασθενής, να είναι ενήμερο, συμφωνούμε όλοι. Τώρα, για την περίληψη. Αυτή η ιδέα της περίληψης πραγματικά είναι προβληματική. Εμείς τι λέμε. Όλες τις πληροφορίες, ε, ενέργειε, ενέργειες, παρενέργειες, ωφέλη και να τα διαβάζει όλα ο ασθενής. Έτσι κι αλλιώς πολλοί δεν διαβάζουν ε, τα χαρτάκια αυτά στα φάρμακα, αλλά εκείνοι που τα διαβάζουν να ξέρουν τι μπορεί να τους προκαλέσει ένα φάρμακο. Εγώ συμφωνώ με την εκτενή ε, πληροφόρηση του φαρμάκου όπως ισχύει σήμερα, όχι περίληψη. Άλλο σημαντικό στοιχείο η ανεξαρτησία. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτή την επιτροπή συμβουλευτική λέγεται εδώ για τη διαχείριση του κινδύνου. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι άλλα πρόσωπα διαφορετικά από εκείνους που συμμετέχουν στον οργανισμό φαρμάκων. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν κάποιος δίδει μια σύσταση, αν συμμετέχει και στην άλλη επιτροπή που θα πρέπει να αξιολογεί τις παρενέργειες, είναι κριτής και κρινόμενος. Τώρα μου λένε ένας από κάθε χώρα. Γιατί δεν πρέπει να είναι συλλογικό το σώμα, δηλαδή ένα συλλογικό σώμα κρατών, ένα συλλογικό σώμα ασθενών, ένα συλλογικό σώμα εμπειρογνωμόνων, όπου να είναι γιατροί ή επαγγελματίες υγείας, σε πάση περιπτώσει. Όχι ένας από κάθε χώρα. Με ποιο κριτήριο θα γίνει αυτό. Υπάρχουν άλλες δομές με συλλογική εκπροσώπηση, πολύ καλή λειτουργία και αξιοπιστία για το σύστημα. Ε, θα πρέπει να ενισχυθεί το κύρος όμως αυτού του θεσμού. Και για τη διαφάνεια, όσο περισσότερη διαφάνεια υπάρχει και πρόσβαση στα δεδομένα, τόσο θα έχουν εμπιστοσύνη στο φάρμακο οι ασθενείς. Και μάλιστα στα νέα φάρμακα και στα φαρμακευτικά εργαστήρια. Αλλά σας παρακαλώ, δεν επιτρέπεται τα εργαστήρια γιατί το είδαμε αυτό στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, α πούμε, για τη γρήπη που είχαμε και συγκρούσει συμφερόντων. Δεν θα πρέπει να διαπλέκονται. Αυτά να είναι ξεκάθαρα ο καθένα στη δουλειά του και έτσι κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι συντονιστές και μόνο που εκτενέστατα αναφέρθηκαν στο θέμα και τώρα παρακαλώ πιο σύντομα οι υπόλοιποι βουλευτές. Η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω τόσο γρήγορα, αλλά όχι σε βαθμό που να μην μπορούν πλέον να με μεταφράζουν οι διερμηνείς. Ε, μελέτησα την έκθεση προσεκτικά και ομολογώ ότι το θέμα είναι δύσκολο τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουμε τον οργανισμό για τα φάρμακα ΕΜΕΑ τα 15 χρόνια με κεντρική αδειοδότηση και από τότε αγωνιζόμαστε για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ε, με μικρή ή καθόλου αποτελεσματικότητα. Η φαρμακοεπαγρύπνηση ή η ασφάλεια ενός φαρμάκου, η γνώση για τα προβλήματα των φαρμάκων είναι ε, τόσο καλή όσο η τροφοδοσία του συστήματος σε πληροφορίες. Και ποιοι είναι αυτοί, τα εθνικά συστήματα υγείας, οι γιατροί, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας. Και θα πρέπει με λιφαλαιότητα να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν το έκαναν οι επαγγελματίες υγείας. Παρόλο που συμφωνώ πάντα με την ε, συντονίστριά μου την κυρία Μακάβαν και συνάδελφο, δεν συμφωνώ στην τροπολογία 3 για τη σύνθεση της Επιτροπής αυτής. Έχουμε μια έκφραση στα γερμανικά που λέει «Βάζω το λύκο να φυλάει τα πρόβατα». Τα κράτη-μέλη εδώ και δέκα χρόνια δεν κούνησαν δαχτυλάκι. Και τι θα βάλουμε τώρα ένα χώρα, ένα μέλος σε αυτή την επιτροπή. Το ότι το θέλουν τα κράτη-μέλη, το καταλαβαίνω αυτό ανθρώπινα, αλλά πολιτικά είναι λάθος. Εργνώμονες, επιστήμονες να στείλουμε εκεί. Όχι εκπροσώπους των οργανώσεων αυτών των εθνικών ε, της υγείας που μέχρι τώρα δεν έχουν σηκώσει το δαχτυλάκι τους δεν έχουν κουνηθεί καθόλου. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό και ε, αντιτίθεται σε ό,τι έχω ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται η Επιτροπή αυτή, η νέα της δομή και λειτουργία, όπως προτείνεται στις τροπολογίες 8 και 9, και πώς συνεργάζεται με την Επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα, το βρίσκω ενδιαφέρον, αλλά δεν είμαι σίγουρη για το πώς λειτουργεί. Έχει δίκιο η κυρία Παρβάνοβα. Ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο. Αφήνω και στην άκρη και άλλα πράγματα, Πρόεδρε, για να μην με διακόψετε και με... Κόψετε. Για την τροπολογία 5, το λεγόμενο μαύρο τρίγωνο. Αν εγώ ήμουν φαρμακευτική εταιρεία, δεν θα έκανα καμία προσπάθεια να βγάλω φάρμακο στην αγορά που να μην έχει περάσει από όλες τις μελέτες. Compassionate use λέγεται αυτό. Ε, πολλοί ε, ασθενείς θέλουν να έχουν φάρμακα πολύ νωρίς. Και μάλιστα ασθενεί με AIDS θέλουν τα φάρμακα αυτά ακόμα και αν δεν έχουν ελεγχθεί πλήρω. Να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν φάρμακα που να μην έχουν περάσει όλα τα στάδια. Το γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα εγώ αν είχα ένα προϊόν με μαύρο τρίγωνο σιγά μην πάρουν και νεκροκεφαλή. Ε, όχι, δεν θα το βγαζα, θα περίμενα να περάσει όλα τα στάδια του ελέγχου για να μην ε, ε πάθει ε, ζημιά η εικόνα μου, η εμπορική και το προφίλ μου. Το είπαν και η κυρία Μακάβαν και η κυρία Παρβάνοβα για τις οδηγίες που είναι μέσα στο φάρμακο. Βεβαίως χρειάζεται καινούρια μορφή γιατί είναι παροχημένη αυτή που κυκλοφορεί σήμερα. Το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δύσκολο. Αλλά γι' αυτό έχουμε φτιάξει και αυτούς τους φορείς. Ε, να... Και εκεί είναι ακριβώς ε, η ε, θέση να γράφει και το κουτί προσοχή, νέο φάρμακο, διαβάστε τις οδηγίες. Τώρα το μαύρο τρίγωνο δεν μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Ja, ein starkes Plädoyer für Wissen. Μάλιστα, περισσότερους επιστήμονες, λιγότερους εθνικούς εκπροσώπους. Ανεξάρτητους επιστήμονες. Αυτό ζήτησες με την ε, αγόρευσή σου. Λίζε, ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Μακάβαν στα περισσότερα θα συμφωνήσω με τα όσα είπε η σκιώδη συγγήτριά μας κυρία Ιούσο. Δύο πράγματα θέλω να παρακαλέσω ωστόσο να σκεφτούμε όλοι μαζί. Αφενός την ανακοίνωση παρενεργειών από πλευρά του ασθενούς απευθεία στις αρχές. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Εάν δεν γίνεται διαφορετικά, αν οι γιατροί ε, τροχοπεδούν και δεν κάνουν την απαραίτητη αυτή εργασία, ίσως τότε πρέπει να ανοίξει αυτή η δυνατότητα αλλά βρίσκω ότι θα είναι ένα αδύναμο σημείο. Κανονικά η σχέση μεταξύ ασθενούς και ιατρού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο ασθενής να μπορεί να ε, συζητεί με τον γιατρό του και ο γιατρός να κοινοποιεί αυτές τις παρενέργειες στις αρμόδιες αρχές. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλοι να σκεφτούμε ποιον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν την υπόθεση. Και εάν βέβαια υπάρχει κατεξαίρεση μια τέτοια περίπτωση όπου ο γιατρός ε, δεν συνεργάζεται, έχει καλώς. Το άλλο τώρα για την ενημερώση των ασθενών, όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, οι πιο ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, άνθρωποι, τους παραπέμπουμε διαρκώς στο διαδίκτυο, αλλά τα φάρμακα τα χρειάζεται ο άνθρωπος κυρίως όταν είναι σε μεγάλη ηλικία και οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν τα πάνε τόσο καλά με το διαδίκτυο. Ένα άλλο θέμα για αυτή την προειδοποίηση με ένα μαύρο κουτάκι. Πολλοί λένε ότι δεν το θέλουν γιατί ε, αυτό το μαύρο περιθώριο ή το κουτάκι ε, στη Γερμανία τουλάχιστον σημαίνει πένθος. Η, το κουτακι στη γερμανια τουλαχιστον σημαινει πενθος ενω τα, τα φάρμακα τα χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε, να σώσουμε τον ασθενή. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται με τρόπο λογικό. Αντιθέτω πάντως με τη γνώμη άλλων συναδέλφων η δική μου δεν είναι ότι θα πρέπει ότι είναι μια λανθασμένη ιδέα η σύνοψη των περισσότερων ιδιωτήτων του φαρμακού. Οι περισσότεροι παρασκευαστές το κάνουν αυτό. Βέβαια γράφουν και ορισμένα πράγματα που τους ε, απαιτούν η νομική του συμβουλή για να μην υφίστανται μεταγωγές, προειδοποίησεις κτλ θα πρέπει να λέει ναι, το, το φάρμακο πρέπει να το πάρετε εφόσον σας το έχει συστήσει ο γιατρός σας και ούτω καθεξής. Άρα όχι μόνο προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί εάν λάβει κανείς το φάρμακο, αλλά και μια προειδοποίηση για το τι θα πάθει ο ασθενής, τι κινδυνεύει να πάθει ο ασθενής, αν δεν ε, λάβει το φάρμακο, αν δεν πάρει το φάρμακό του ή αν δεν το πάρει με τον σωστό ενδεδειγμένο τρόπο. Επίσης τι πρέπει να κάνει εάν συμβεί κάτι, ότι πρέπει να το συζητήσει με τον γιατρό του. Εγώ τα είδα τα πρότυπα αυτά, τα βρίσκω πολύ καλά. Γνωρίζω ότι τα χαρτάκια με τις οδηγίες δεν είναι πάντοτε διαυγή ούτε για τους γιατρούς ούτε για τους ασθενείς. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πετάξουμε αμέσως ε, το έγγραφο της Επιτροπής, αλλά να τη το ζητήσουμε ήδη από σήμερα να τα διατυπώσει ακριβέστερα. Διότι ποια είναι για παράδειγμα μια χαρακτηριστική ιδιότητα ενός φαρμάκου. Ο καθένας αν δεν το διατυπώσουμε ακριβέστερα θα έχει διαφορετική άποψη. Ίσως λοιπόν μπορεί να το διατυπώσει ακριβέστερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως προς την κατεύθυνση που είπα εγώ, διότι ο καθένας αλλιώς θα βάλει τη δική του ερμηνεία και το μόνο που κάνουμε είναι με την, στην περίπτωση αυτή να απασχολούμε περισσότερο τους δικηγόρους. Ενώ αυτό που θέλουμε είναι η καλύτερη μεταχείριση του ασθενούς. Ευχαριστώ. Ούλμερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια. Η φάρμακο επιτήρηση είναι σημαντικό θέμα. Ας μην λησμονούμε ότι καμιά φορά είναι και αυθαίρετος χαρακτηρισμός ενεργειών και παρενεργειών. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια βελτιωμένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων και ακριβώς εάν οι χώρες μέλη συμμετάσχουν πλέον σε ένα όργανο, αυτό θα παρεμποδιστεί να γίνει. Ενώ αυτό που χρειάζεται είναι μια επανεξεργασία της τράπεζα αυτής δεδομένων με τρόπο επιστημονικό. Έχω και ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία θα εξοπλίσω και με τροπολογίε. Θα πρέπει να δοθούν δυνατότητες και όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, αλλά και με φάξ ή με άλλου τρόπου να μπορούν να ενημερώνονται οι άνθρωποι και τι γίνεται και με τους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν τα φάρμακα αυτά ως soft label use, δηλαδή όχι ακριβώς όπως τα ε, γράφει ο γιατρός στη συνταγή, αλλά και για ε, θεραπεία άλλων συμπτωμάτων ή νόσων. Για μένα τίθεται επίση το ερώτημα, μπορεί ο ασθενής να έρθει κατευθείαν σε επαφή με την αρμόδια αρχή, για παράδειγμα στέλνοντα ένα φαξ και να ξεκινήσει έτσι τότε αυτή την περίπλοκη διαδικασία. Ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Ένα ασθενή. Κάτι που είναι σύνηθε στη Γερμανία. Επειδή δίνουν συχνά τα φαρμακεία τα generic δηλαδή αυτά τα χωρίς ε, εμπορική επωνυμία και πει ο ασθενής κοιτάξτε το φάρμακο που μου έδωσε το φαρμακείο αντί για αυτό που είχε γράψει ο γιατρός και υποτίθεται ότι είναι ε, η ίδια ενεργός ουσία, μου μυρίζει διαφορετικά. Γράφω ένα φάξ και το στέλνω στην αρμόδια αρχή. Τι θα γίνει τότε. Έχω λοιπόν ότι αυτό θα έχει χαρακτήρα αποτρεπτικό. Γνωρίζουμε ότι ένα τρίτο περίπου των ασθενών δεν παίρνει καν τα φάρμακα. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει και τα αγοράζει από το φαρμακείο. Εν πάση περιπτώσει, εν το συνόλο του νομίζω ότι η έκθεση είναι καλή, αλλά πρέπει τα συστήματα που θα προτείνουμε να είναι ξεκάθαρα, οι γιατροί να είναι διατεθειμένοι να κάνουν τις σχετικές κοινοποιήσεις στις, στις αρμόδιες αρχές για τις περίπτωσεις παρενέργειων των φαρμάκων και το καθεξής. Το φάρμακο μυρίζει διαφορετικά, λέτε, και γι' αυτό ε, στέλνει το φάξ. <laughs> Άρα δεν είναι η γεύση που τον ενοχλεί τόσο πολύ. Ενδιαφέρον το παράδειγμα. Ο κ. Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Μακέβαν για το καλά δουλεμένο κείμενο, το σχέδιο έκθεσης, αλλά και τη συνάδελφό μου την κυρία Ριβασή για τον εκτενή σχολιασμό και τις τροπολογίες που ε, προσυπογράφω επίσης. Θα ήθελα όσο πιο σύντομα γίνεται να εστιάσω σε δύο σημεία. Ε, το πρώτο, αυτό που έχω αναφέρει και άλλη φορά σε αυτή την αίθουσα, είναι ότι οι αρμοδιότητες για την φαρμακοεπαγρύπνηση και τα φαρμακευτικά νομοσχέδια ε, μεταφέρθηκαν από τη διεύθυνση που είχε ως κύριο ε, μέλημά της την υπεράσπιση των συμφερόντων της βιομηχανίας και των κερδών της σε μια διεύθυνση της Επιτροπής που εστιάζει στη δημόσια υγεία και το συλλογικό συμφέρον. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι στο παρόνομο σχέδιο υποβόσκει μια τάση να εισάγονται επισπεσμένα φάρμακα στην αγορά χωρίς ε, ενδελεχείς κλινικές δοκιμές και με συνοπτικές διαδικασίες αδειοδότησης με το σκεπτικό ότι θα υπάρχει ένα ενδυναμωμένο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, ανάλυσης των κινδύνων και αναφοράς των ανεπιθύμητων παρενεργειών των ε, φαρμάκων. Αυτό εμάς μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Και αφουγκραζόμαστε την κοινωνία των πολιτών και την οργανωμένη της έκφραση. Ζητάμε πιο αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης πριν ένα φάρμακο μπει στην αγορά ταυτόχρονα με την παράθεση των αποτελεσμάτων συγκριτικών κλινικών δοκιμών αλλά και την απόδειξη της ε, προστιθέμενης θεραπευτικής του αξίας. Είναι φανερό ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τους πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από ένα νέο φάρμακο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους και να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο συντονιστικό όργανο των Εθνικών Επιτροπών Φαρμακοεπαγρύπνησης. Το σύστημα αναφοράς και παρακολούθησης των ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων πρέπει να παραμείνει υπό την επίβλεψη των δημόσιων αρχών. Ενώ πρέπει να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη, τον ασθενή συγκεκριμένη περίπτωση, σύστημα αναφορών προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρείε πολλές φορές αποκρύπτουν, όπως ήδη έχει αναφερθεί, τις ανεπιθύμητες παρενέργειες ή τις δημοσιοποιούν όταν είναι αργά με σημαντική χρονική καθυστέρηση. Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που συζητάμε, η Ondra Vigilance, πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη και να είναι εύκολα προσβάσιμη από το κοινό, το οποίο πρέπει να είναι πολύ καλά πληροφορημένο για τις δυνατότητες αναφοράς των ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλω να σταθώ σύντομα είναι το θέμα των περιβαλλοντικών ε, επιπτώσεων και των κινδύνων των φαρμακευτικών προϊόντων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διοργάνωσε πέρσι ένα σεμινάριο εμπειρογνωμόνων για τα φαρμακευτικά προϊόντα και δημοσίευσε μόλις στις 13 Ιανουαρίου τα συμπεράσματα της συνάντησης μέσω μιας τεχνικής έκθεσης. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι διαδικασίες για την έγκριση των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίρνουν υπόψη τους τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εγκυμονούν τα εν λόγω προϊόντα. Επιπλέον, καλεί για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα ότι πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους ως προς το περιβάλλον και για τα προγράμματα ανάκλησης φαρμάκων ότι πρέπει αυτά να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώνεται επίσης στην έκθεση ότι τα φαρμακευτικά απόβλητα θα πρέπει πάντα να αποτεφρώνονται. Η Επιτροπή μέσω της φαρμακοεπαγρύπνησης θα έπρεπε να δώσει συνέχεια σε αυτά τα πορίσματα της έκθεσης που αναφέραμε, είτε έμεσα είτε άμεσα, κυρίως με το να θεσμοθετήσει την υποχρέωση να παρακολουθούνται και να αναφέρονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και να συγκρίνονται αυτά τα δεδομένα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που παρουσιάζουν οι εταιρείε κατά τη διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης των νέων φαρμάκων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα περιφερειακά και τα εθνικά κέντρα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να ενδυναμωθούν και να εναρμονιστούν με τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, αλλά και να διασυνδεθούν διαδικτυακά με αυτήν, ώστε να παρέχουν διαφανή και αξιόπιστα δεδομένα στους χρήστες, δηλαδή τους ασθενείς, τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια που επεξεργάστηκε ένα θέμα δύσκολο και που πάντως χρειάζεται να λυθεί γρήγορα. Συμφωνώ όπως και η κυρία Ροτ Πέρεντ ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να συνδεθεί, να απαρτιστεί από εκπροσώπους των χωρών μερών. Εδώ χρειάζεται να είναι επιστήμονες. Εάν τώρα είναι και κάποιοι επιστήμονες από κάποια χώρα μέρο, εντάξει, αλλά όχι όμως να καθοριστεί από τώρα σε ποιες χώρες, από ποιες χώρες θα εκπροσωπούνται ε, όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την επιτροπή. Τώρα, όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι μια τράπεζα δεδομένων ευρωπαϊκή, διότι μόνο εκεί μπορεί να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα λαμβάνει τις πληροφορίες η τράπεζα δεδομένων. Θα βάλουμε και τους ασθενείς μέσα, εντάξει. Αυτό είναι μια δυνατότητα. Αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις. Εάν δώσουμε μόνο στον ασθενή την πληροφορία, νομίζω ότι η πληροφορία μπορεί να λάβει σοβαρό χαρακτήρα μόνο εφόσον συζητηθεί με τον γιατρό, ο οποίος ε, έχει γράψει τη συνταγή, ή με τον φαρμακοποιό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βάλουμε εδώ κάποιον φραγμό, ώστε να μην εμφανίζονται και κάποιες ε, προειδοποίησεις ας πούμε χαρακτήρα λαϊκιστικού. Για παράδειγμα με το συμβόλιο, με το εμβόλιο της, ε, του αυτόδου πυρετού των χείρων που τίθεται ότι πέθαναν και άνθρωποι επειδή ε, κάπως ε, πέρασε αυτό ε, στον ανθρώπινο οργανισμό. Να δούμε λοιπόν, να σκεφτούμε με ποιον τρόπο θα, θα τροφοδοτείται η, η ε, τράπεζα δεδομένων με πληροφορίες. Τώρα, για το φυλάδιο που ε, μπαίνει μέσα στο κουτί του φαρμάκου. Αυτό που πρωτίστως με ενδιαφέρει εμένα όταν θέλω να πάρω ένα φάρμακο είναι η δοσολογία που χρειάζεται καμιά φορά να ψάχνω πολύ μέχρι να την βρω μέσα στο φυλάδιο. Αυτό το μαύρο τρίγωνο και εμένα μου φαίνεται μάλλον απορριπταίο. Σίγουρα μπορούμε να το υιοθετήσουμε αλλά μπορεί και να οδηγήσει στο ότι ο ασθενής που ε, του έγραψε ο γιατρός ένα φάρμακο, άπαπα βλέπω πάνω το μαύρο τριγούνο, δεν το παίρνω το φάρμακο. Άρα ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις πληροφορίες που δίνουμε. Νομίζω ότι οι πληροφορίες πρέπει να μπαίνουν στο φυλάδι αυτό, στο χαρτάκι αυτό και οι πληροφορίες μέσω διαδικτύου μόνο μου φαίνεται ότι δεν είναι χρήσιμο. Πολλοί που έχουν ανάγκη από τι υποχρεώσει αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Άρα χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Φαξ ή επιστολή. Ακόμα και οι γιατροί καμιά φορά δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα. Σας ευχαριστώ. Καρλ Σλούτερ τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όμως, παρόλα αυτά, έχω και εγώ τις παρατηρήσεις μου. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μακάβανη, η οποία προχώρησε πολύ σε πολλά ζητήματα. Αλλά να σας πω το εξής σήμερα όποιος είναι θύμα παρενέργειας ενός φαρμάκου έχει την τάση να παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο στα νούμερα που εμφανίζονται στο χαρτάκι που συνοδεύει τα φάρμακα με τις ενδείξεις και τις οδηγίες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι οι κατάλληλες πληροφορίες φτάνουν στα χέρια των κατάλληλων προσώπων τελικά. Και από την πλευρά του Κοινοβουλίου μην ξεχνάμε ότι ανέκαθεν αγωνιζόμαστε για να υπάρχει επαρκή ενημέρωση για τι παρενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια και στο θέμα αυτό. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα με το μαύρο τριγωνάκι, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το τριγωνάκι αυτό, υπάρχει και σχετικός Το μαύρο τρίγωνο δεν έχει κανένα σκοπό να αποκρύψει τίποτα από τον καταναλωτή, Σε αυτό το διατηρήσουμε εφόσον από τη στιγμή που συνταγογραφείται ένα φάρμακο δεν θέλουμε να παραμείνει στη βάση δεδομένων εάν έχει αδειοδοτηθεί αλλά και όχι. Δηλαδή, όταν κανεί παίρνει ένα φάρμακο με μαύρο τριγωνάκι, είναι πιο προσεκτικό σε σχέση με τι ε, παρενέργειε και μπορεί να τι παρακολουθήσει και καλύτερα. Γιατί καμιά φορά οι παρενέργειες μπορεί να είναι και πιο σοβαρέ από αυτό που φανταζόταν κανεί, αλλά μπορεί και λιγότερο. Οπότε σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να μπορεί κανεί να αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση που εμφανιστούν. Μπορεί να πρέπει να απαγορευτεί άμεσα ένα φάρμακο εάν έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει τέτοια ανησυχία με το μαύρο τριγωνάκι. Επίση, δεν καταλαβαίνω ακριβώ. Γιατί όλες αυτές οι παρενέργειες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στις οδηγίες χρήσης του φαρμάκου. Θα ήταν ενδιαφέρον κάποιες να αναφέρονται, όπως συνήθως, οι, οι πιο συνηθισμένες ή λιγότερο συνηθισμένες, λόγω χάρη το να πάρει κανείς ένα καταπαρεντικό να δει ότι μπορεί να προκαλέσει αυτό ρεθισμό στο δέρμα. Ε, ε, εγώ αντιλήφθηκα από τη λήψη ενός τέτοιου φαρμάκου ο ίδιος ότι μια τέ, ένας τέτοιος αριθμός στο δέρμα που ο ίδιος ε, είχα μετά από τη λήψη ενός τέτοιου φαρμάκου δεν με ανησύχησε καθόλου τελικά, δεν ήταν τόσο σοβαρή και το γεγονός ότι είχα ενημερωθεί γι' αυτό με έκανε ίσα ίσα να είμαι πιο ήσυχος θα πρέπει λοιπόν οι ενδείξει να επιτρέπουν στου ανθρώπου να είναι πιο ήρεμοι σε σχέση με τη λήψη φαρμάκων, αλλά να αντιδρούν και πιο γρήγορα εφόσον αυτό χρειαστεί. Πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτό είναι ο βασικό μα στόχο. Και ολοκληρώνοντα ω προ την προστασία του περιβάλλοντο, δεν έχουμε νομίζω σταθεί επαρκώ στο θέμα αυτό. Στη Σουηδία υπάρχει ένα σύστημα που επιτρέπει την ταξινόμηση των ε, ε, επιπτώσεων για το περιβάλλον σε τέσσερι βαθμίδες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Έτσι υπάρχουν τρία επίπεδα πληροφόρησης. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πληροφόρηση του ασθενούς και αυτή στιγμή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει ο ασθενής να φροντίσει να αντιδράσει άμεσα. Επίσης υπάρχει πληροφόρηση προς τον φαρμακοποιό και μετά η πληροφόρηση προς τους ε, ειδικούς της υγείας. Πληροφορίες που προσαρμόζονται ανάλογα με το ποιο είναι ο παραλήπτη των πληροφοριών. Νομίζω ότι ο τρόπος αυτός είναι αρκετά καλός και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε τους γεωργού τους ηχθειοτρόφους, οι οποίοι και αυτοί μπορεί να χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε περισσότερο στο ζήτημα αυτό, διότι η συνέπειση των περιβάλλων είναι στοιχείο σημαντικό Υπάρχουν αρκετά προβλήματα σήμερα, τα οποία σχετίζονται ακριβώ με την υπερβολική χρήση κάποιων φαρμάκων. Ευχαριστώ. ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να λάβετε θέση, παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα την εισηγήτρια για την συνεργασία. Ευχαριστώ για τα πολλά θετικά σχόλια για την πρότασή μας. Παρόλες τις συζητήσεις που έγιναν, διαπιστώνω ότι επί ουσιοδών θεμάτων δίνεται μεγάλη υποστήριξη στις προτάσεις της Κομισιόν και στο σχέδιο εκθέσεως, κυρίως για το θέμα της ε, Κεντρικής Τράπεζας Δεδομένων, της Ultra Vigilance, της ε, Periodic Safety Report, και patient reporting, λέω μόνο λίγα παραδείγματα. Η εισηγήτρια συνιστά σε ορισμένα από τα θέματα αυτά να κάνουμε πιο θαραλία βήματα από αυτά που ίσως ε, πρόβλεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της. Για μας θα είναι δύσκολο βέβαια να αντιταχθούμε σε τροπολογίες οι οποίες θα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση όπως η πρότασή μας, και ενισχύουν κάποια στοιχεία τους, για παράδειγμα την διαφάνεια, την ε, διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων, όπου εμείς δεν προχωρήσαμε τόσο πολύ όσο τώρα το σχέδιο εκθέσεως. Αλλά νομίζω ότι κατά βάση όντως κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση και η περαιτέρω διαδικασία θα μπορέσει να εξελιχθεί χωρίς ε, δυσκολίες και να καταλήξει σε θετική έκβαση. Κάτι που φαίνεται να είναι πλέον αμφιλογόμενο είναι, για παράδειγμα πρώτο, η σύνθεση της Επιτροπής, του Κομιτέ, της Επιστημονικής Επιτροπής. Στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου συζητήσαμε το θέμα αυτό ήδη για αρκετό καιρό. Το βασικό επιχείρημα των χωρών μελών είναι αυτό της επικοινωνίας του κινδύνου. Να υπάρχει μία φωνή σε κάθε χώρα μέλος που να μπορεί να ενημερώνει την κοινή γνώμη για του κινδύνου των φαρμάκων που κυκλοφορούν. Αυτό βέβαια είναι αντίθετο με την πρότασή μα. Από την άλλη μεριά έχουμε κάποια κατανόηση. Αλλά βέβαια δεν είναι και το μοναδικό στοιχείο τη πρότασή μα. Στην πρότασή μα, για παράδειγμα, προβλέπουμε και επιλογή μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, του Management Board και όχι μόνο της χώρας μέλους. Και υπάρχει κάποια διασύνδεση και με τον ρόλο της Επιτροπής. Στο σχέδιο εκθέσεως είδαμε ότι ζητείται αναβάθμιση της Επιτροπής και αυτό το θεωρούμε σωστό. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η σχέση της φαρμακοεπαγρύπνησης και της Επιτροπής που ασχολείται με φάρμακα για νόσους ανθρώπων στην, ε, στον, στην οργάνωση, όπου όμως, εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή είναι εκείνη η οποία έχει τον τελευταίο λόγο και σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν και σύμφωνα με την πρόταση της εισηγητρία σας. Αυτόν τον αναβαθμισμένο ρόλο της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης εμείς τον ορώμεθα θετικά και θεωρούμε ότι αυτό προσφέρει και μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην κρίση σχετικά με ανεπιθύμητες παρενέργειες. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπέρ του αναβαθμισμένου ρόλου της Επιτροπής Φάρμακο Επαγρύπνησης. Έρχομαι τώρα στο φυλάδιο που χορηγείται μαζί με το φάρμακο, στο ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνεται πάντοτε στα κουτιά των φαρμάκων. Νομίζω ότι τον Μάιο του 2007 παρουσία του Επιτρόπου Φερχόγγεν ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν προτάσεις για βελτίωση του σημειώματος αυτού που συνοδεύει τα φάρμακα. Το θέμα είναι δύσκολο. Στην ανακοίνωσή μας προτείναμε να συνοψιστούν οι παρενέργειες κυρίως αυτές που έχουν μεγαλύτερη συχνότητα και είναι και πιο σημαντικές. Τότε βέβαια επικριθήκαμε ότι στην σύνοψη αυτή βάζουμε μόνο τις παρενέργειες και μας ζητήθηκε να βάλουμε και τις θετικές και τις αρνητικές ας πούμε παρενέργειες στην σύνοψη αυτή. Και γι' αυτό προτείναμε τώρα αυτήν την σύνοψη και απαντώντας τον κύριο Λίζε υποτίθεται ότι θα, αναφέρονται και τα θετικά αποτελέσματα και τα αρνητικά αποτελέσματα και κυρίως τα πιο συχνά και τα πιο σημαντικά. Γιατί συχνά ο ασθενής σήμερα δεν το διαβάζει όλο το σημείωμα. Έχουμε άλλωστε υποστήγη και κριτική για την πρότασή μας αυτή, το γνωρίζουμε νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα βήμα προς τα εμπρός στην περαιτέρω διαδικασία και εν προκειμένου ε, προς το συμφέρον πάντοτε του ασθενούς. Θα έρθω τώρα σε ορισμένα σημεία κριτικής. Πρώτα για τη χρηματοδότηση. Ήδη τώρα έχουμε καθυστερήσεις με την ίδρυση της Τράπεζας Δεδομένων για την φαρμακοεπαγρύπνηση που οφείλεται εν μέρη και στα δημοσιονομικά, στον προπολογισμό. Η τράπεζα αυτή είναι αυτή που καταβροχθίζει και τα περισσότερα κονδύλια από όλε τι τράπεζε δεδομένων. Δεν θα πω τώρα στι εσωτερικέ συζητήσει τη Κομισιόν, αλλά η community subvention εδώ δεν έχει αυξηθεί. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η βιομηχανία δεν συμμετέχει στο, συμβούλιο, εποπτικό συμβούλιο, ούτε σε κανένα άλλο όργανο το οποίο πρόκειται να ε, συζητήσει ή να αποφασίσει σχετικά με την ultra vigilance στο μέλλον. Πολύ περισσότερη είναι η επιρροή της ε, βιομηχανίας για την έγκριση του φαρμάκου και πολύ λιγότερη για τα μετά την έγκριση, αδειοδότηση δηλαδή. Το άλλο τώρα, για το earlier approval, ότι με την πρότασή μας δηλαδή θέλουμε να προωθήσουμε ταχύτερα τα φάρμακα προς την έγκρισή τους. Σας λέω καθαρά ότι όχι στην νομοθεσία μας διαθέτουμε μέσα που μας επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις ε, να δίνονται οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των φαρμάκων νωρίτερα, για παράδειγμα για πολύ σπάνιες νόσους, αλλά αυτά όμως είναι συγκεκριμένα και κατ' εξαίρεση. Με κανένα τρόπο δεν θέλουμε να αλλάξουμε εδώ την ισορροπία. Σας το εγγυώμαι. Ολοκληρώνοντας, ατενίζουμε την περαιτέρω διαδικασία με αυτοπεποίθηση. Η Κομισιόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μεταβατική περίοδο. Όμως ο ίδιος ο υποψήφιος επίτροπος Νταλή είπε και στην ακροασία του εδώ ενώπιόν σας ότι ενδιαφέρεται και στο θέμα αυτό να προχωρήσει γρήγορα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κινηθούμε όντως προς την κατεύθυνση αυτή και να παραγάγουμε αποτελέσματα σύντομα. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που δώσατε σε σημαντικά σημεία της προτασεώς μας. Σας ευχαριστώ και Τίερ Μπέργκερ για την παρέμβασή σας. Θα ακολουθήσει η συγγήτρια, η οποία έχει ακόμη να πει κάτι στο τέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και για την προσοχή και τη φροντίδα που δείχνουν ε, για το θέμα αυτό. Ο καθένας θέλει να είναι όσο γίνεται καλύτερο το σύστημα. Μπορεί να έχουμε επιμέρους διαφωνίες μικρές, αλλά όχι στο ουσιαστικό θέμα και την επιθυμία μας να βοηθήσουμε. Ε, για την Επιτροπή αυτή και ποιος συμμετέχει. Στην αρχή συμφωνούσα με την Dagmar, γιατί και έχω πάει και εγώ στον Οργανισμό Φαρμάκων, στην ΕΜΕΑ και ξέρω τι δυσκολίες υπάρχουν. Και έλεγα να είναι επιστήμονες, ναι. Αλλά μετά άκουσα και το Συμβούλιο και το ε, ΕΜΕΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατάλαβα. Γιατί ορισμένοι ε, επιστήμονες θα είναι από τις εθνικές αρχές. Δεν θα είναι οποιοδήποτε πρόσωπος εθνικός, θα είναι επιστήμονες και από τους οργανισμούς φαρμάκων. Έξι μήνες μόνο αυτό το θέμα συζητούσε το Συμβούλιο, που αφήστε που δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο σημαντικότερο. Εμένα με σόκαρε ότι μετά από έξι μήνες, τρεις, τέσσερις ομάδες εργασίας να συζητάνε μόνο αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να συζητούν το άλλο που είναι πολύ σημαντικότερο. Εντάξει. Θα μπορούσα να το δεχτώ αυτό, να συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι αυτοί όλων των κρατών μελών. Βεβαίως να είναι άνθρωποι ικανοί, ανεξάρτητοι που να εργάζονται προς ε, όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί το είπα αυτό, γιατί το πρότεινε δίνουμε πιο εξέχοντα ρόλο σε αυτή την Επιτροπή. Γιατί σήμερα τι συμβαίνει και το συζήτησα αυτό με την ΕΜΕΑ. Επειδή δεν έχει καμία εξουσία σήμερα η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης παρά μόνο κάποιες ασαφείς ε, συστάσεις και θολές κάνει, δεν λειτουργεί σωστά. Για να λειτουργεί σωστά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει επίσημα συστάσεις. Ε, Βεβαίως η Επιτροπή για τα Φάρμακα θα παίρνει την τελική απόφαση, αλλά δεν θα μπορεί να ανατρέπει την ε, θέση της νομοδοτούσας επιτροπής. Τώρα αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σκοπός είναι να είναι μια σωστά λειτουργούσα επιτροπή και να μην πηγαίνουν εκεί κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι ε, για να αναφέρουν στοιχεία αριθμητικά και στατιστικά, αλλά κάποιοι επιστήμονες με γνώσεις και με ε, εργασία σε αυτό το θέμα. Ε, για την άμεση προφόρηση των ασθενών, το είχα ξανασυζητήσει αυτό. Δεν συμφωνώ να πηγαίνουν στην ΕΜΕΑ και να ρωτούν οι ενδιαφερόμενοι για τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Σούλμερ. Χρειάζεται ένα φίλτρο στην Εθνική Αρχή που να διηθεί ε, σε χώρες που υπάρχουν οι δηλώσεις των ασθενών δεν ε, καταγράφουμε ό,τι μας λένε οι ασθενείς. Έχουν το όνομα του ασθενούς, το τσεκάρουν, το ελέγχουν, κοιτούν, επαληθεύουν αν είναι πραγματική πληροφόρηση και μετά ε, το δηλώνουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Δεν είναι ο καθένας που έχει τον πόνο του να πηγαίνει να τον λέει στην Επιτροπή και γι' αυτό να παραμένει ε, ως φίλτρο ο εθνικός οργανισμός. Γιατί στην ΕΜΕ αυτό που θα σας πούνε ότι το τελικό αποτέλεσμα ε, είναι τόσο καλό όσο ε, είναι αυτό που τροφοδοτεί. Δηλαδή άμα βάλετε βλακίες, βλακίες θα βγουν και στο τέλος. Για το τρίγωνο, εγώ δεν έχω καμία αιμονή με τρίγωνα ή άλλα σύμβολα. Για το τρίγωνο που προτείνω είναι ήδη στο φυλάδι οδηγιών για ε, τους ασθενείς, όχι πάνω στο ε, κουτί. Εγώ δεν είμαι επαγγελματία υγείας εδώ, πολλοί από εσά είστε. Είναι ένα αναγνωρισμένο σύμβολο στην υγεία ε, ως ένα προϊόν που ελέγχεται στενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να έχουμε τρίγωνο στο σημείωμα γύρω-γύρω αστερίσκους. Δηλαδή για να δώσουμε νέα πληροφορία για ε, τα χάπια. Μα αυτό το τρίγωνο υπάρχει ήδη και το αναγνωρίζουν ως κάτι συγκεκριμένο. Ήδη οι επαγγελματίες υγείας, μην τους περδέψουμε περισσότερο. Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, εντάξει. Εγώ δεν έχω έμονη ιδέα, ούτε επιμένω για το τρίγωνο, αλλά να γνωρίζουν οι ασθενείς τι παίρνουν, τι είναι αυτό το φάρμακο. για το φυλάδιο το ενημερωτικό, το φύλλο οδηγιών που συνοδεύει τα φάρμακα στο κουτί, θα πρέπει να παραμείνει βασική πληροφορία. Πώς θα το κάνουμε αυτό με περίληψη, δεν ξέρω, χρειάζεται ακόμα συζήτηση. Και ένα τελευταίο. Α, χαίρομαι που το έλυσε αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ξεκαθάρισε ότι μέσω της πρότασης αυτής ε, μπορεί να υπάρχει το παραθυράκι της ταχύτερης αδειοδότησης του ε, φαρμάκου το συζήτησα, το κοίταξα, το μελέτησα, το κατάλαβα και πάλι δεν είμαι ειδική της υγείας. Δεν ε, έχει καμία σχέση αυτό με το ρυθμό χορήγησης της άδεια και της διαδικασίας. Είναι ξεχωριστή η διαδικασία και χαίρομαι που το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ξεκαθάρισε. Και τέλος, ε, όλα αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα που ανέφερε ο συνάδελφος ε, ο Πράσινος και ο Κάρλ τι κάνουμε με το νερό και τα λοιπά. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα πρέπει να μπει σε αυτή την νομοθεσία. Δεν ξέρω πού θα μπει. Υπάρχουν άλλοι που είναι παλαιότερα μέλη εδώ, ίσως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός ο αντίκτυπος για το περιβάλλον δεν ξέρω πού μπορεί να μπει. Εδώ δεν το βλέπω να έχει θέση. Αυτά προς το παρόν και προσβλέπω ε, στις τροπολογίες σας για αποτελεσματική συνεργασία. Ευχαριστώ την εισηγητρία και όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εντατική αυτή και εκτενή συζήτηση. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 3η Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Και... Μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε ψηφίσει κιόλας στην Επιτροπή μας. Και πάμε στο τελευταίο για σήμερα θέμα, εξίσου σημαντικό, ψευδεπίγραφα φάρμακα, τροποποίηση της οδηγίας τάδε, που ισχύει σήμερα και η συγγήτρια είναι η κυρία Μαρίσα Ματίας και της δίνω αμέσω το λόγο. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι για αυτή την πρόταση της Κομισιόν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα που αποσχολεί όλο και περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες αυτή τη διάσταση να μην την ξεχνάμε. Η δική μου βασική μέρημνα ήταν ε, να προσπαθήσω να διασφαλίσω το κοινό συμφέρον σε έναν τομέα, σε έναν χώρο, όπου υπάρχουν πολλά αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα. Σίγουρα διαφορετικά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της έκθεσης που προσπάθησα να συντάξω. Εδώ ήθελα να παραθέσω τα λόγια του κυρίου Φερχόγγεν σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από ένα μήνα περίπου, σε μια γερμανική εφημερίδα, Die Welt, και για να μην μεταφράζω τα λεγόμενα του Επιτρόπου, που ούτως ή άλλως είναι το μεταφρασμένο τμήμα μιας συνέντευξης ε, από τα αγγλικά, θα σας τα διαβάσω κατευθείαν στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Έλεγε λοιπόν ο Επίτροπος Φερχόγγεν ότι ο όγκος των παρεποιημένων φαρμάκων στην Ένωση συνεχώς διωγγώνεται και στο φάσμα και στον ίδιο τον όγκο και ότι οι εμπειρογνώμονες είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το φαινόμενο αυτό. Πριν από δύο μόλις μήνες, 34 εκατομμύρια παραπημένα φάρμακα κατασχέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω στοχευμένων σημείων στα κράτη-μέλη. Ο Επίτροπος λέει ότι αυτό είχε ξεπεράσει τους χειρότερους φόβους μας. Μιλάμε κυρίως για αντιβιωτικά, για φάρμακα κατά του καρκίνου, της ελονοσίας, τα οποία πρόκειται βεβαίω να, τιμωρηθούν, για τα οποία πρόκειται να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι κατά τον πιο αυστηρό τρόπο. Τέλο του παραθέματο. Βάσει αυτή του παραθέματο, λοιπόν, τη συνέντευξη του Επιτρόπου Φερχόγγεν, ε, είναι μια αφορμή καλή αυτή για να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο για το έργο του ω τώρα. Για την καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμάκων αλλά νομίζω ότι η κατάσταση αυτή ακριβώς θέτει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οδηγία και την τροποποίηση μιας οδηγίας που θα πρέπει να μας αναγκάσει να αντιμετωπίσουμε το σύστημα διανομής των φαρμάκων και συγκεκριμένα των παραποιημένων. Εγώ από πλευρά μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για, την... για το σκοπό αυτό, το συγκεκριμένο δηλαδή σκοπό προστασίας των ασθενών. Τώρα, έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή, μπορούμε να εξετάσουμε την έκθεση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω απευθείας όλους, αμέσως μάλλον όλους τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα σταθώ σε όλα τα σημεία της πρότασής μου, ούτε της έκθεσης, ε, όπως φαντάζεστε. Ήθελα απλώς, συνάδελφοι, να σταθώ σε μερικά από τα σημαντικότερα κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη. για τη συζήτηση δηλαδή που έχουμε εδώ. Σημεία για τα οποία έχω ιδιαίτερη περιέργεια να ακούσω τα σχόλιά σας και τα επικριτικά και τις προτάσεις σας. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση δεν ήθελα να επεκταθώ ιδιαίτερος, θα έχετε και άλλες ευκαιρίες να σχολιάσετε. Κάτι λοιπόν που έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά όλη μας συζήτηση, η νομική βάση. Η Επιτροπή στέκεται ιδίω στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φαρμάκων και κυρίως τα θέματα προστασίας των ασθενών. Αυτό είναι και το κέντρο του προβλήματος και του προβληματισμού μας. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα μπορούν να βλάψουν σοβαρά τους ασθενείς είτε λόγω της έλλειψης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων που αναμένονται, είτε λόγω εγγενών ελαττωμάτων των φαρμάκων που γίνονται αντικείμενο εμπορία. Ήθελα λοιπόν να σταθώ και σε αυτό το σημείο ξανά. Τώρα, κάποιες προσθήκες που έκανα στην πρόταση της Επιτροπής. Πρέπει να είναι σαφές ότι στους ορισμούς για να μην πάμε σε μια πιο περίπλοκη και λιγότερο εύληπτη πρόταση, αλλά για να κάνουμε ακριβώς την εντύπωσή μας πιο διαφανή και πιο κατανοητή, να είναι κατανοητό αμέσως για το τι μιλάμε, να σκεφτούμε εδώ λόγου χάρη την αλυσίδα διανομής. Γιατί δυνατότητε δυνατότητες έχουμε για αυτή τη διανομή. Εδώ έχουν προσθεθεί κάποιοι ορισμοί, όπως το ψευδεπίγραφο ε, φάρμακο, το δραστικό συστατικό, τους φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα διανομής και γίνονται και κάποιες διακρίσεις μεταξύ λόγου χάρη των πρακτόρων και των, μάλλον των μεταφορέων και των εμπορευομένων. Πιστεύω ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να προλάβει την σύγχυση και να μην αφήσει κανένα περιθώριο ώστε να παραμένουν γκρίζες περιοχές, γκρίζες ζώνες. Θα πρέπει στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών και της παραπίσης των φαρμάκων να είμαστε αυστηροί. Ορισμοί λοιπόν πιο εύστοχοι, πιο ξεκάθαροι, απλούστεροι και περισσότερο κατανοητοί. Σημείο τώρα, το σημείο που αφορά τους κανονισμούς ασφαλείας. Πιστεύω ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για τα φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται. Είναι αντικείμενο ιατρικής συνταγής. Εδώ πάλι γίνεται μια διάκριση. Διότι νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα για τα προβλήματα που πιο άμεσα μας απασχολούν. Γνωρίζω επακριβώς ότι παραποίηση και αλλίωση φαρμάκων μπορεί να αφορούν και γενώσιμα αλλά και φάρμακα συγκεκριμένη μάρκας. Το θέμα λοιπόν είναι και το κόστος των προϊόντων και το τι κέρδος μπορεί να αποκομίσει κανείς από την παραποίηση συγκεκριμένων ε, προϊόντων, φαρμάκων. Και αυτό γενικεύει βεβαίω το πρόβλημα σε πολλέ περιπτώσει. Υπάρχει λιγότερο κέρδο όταν παραποιείται ένα γενώσιμο φάρμακο, μάλιστα, επειδή ακριβώ είναι χαμηλό το κόστο των φαρμάκων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν τα μέτρα ασφάλεια, το σύστημα ασφάλεια πρέπει να είναι υποχρεωτικό και αυστηρό. Ιδίω για τα γενώσιμα φάρμακα. Όπω λέει και η Κομισιόν πρέπει να γίνει μέσω μια ανάλυση κινδύνων. Γνωρίζω ότι πολλοί από τους κοιόδης εισηγητές ε, θέλουν μέτρα ασφαλείας υποχρεωτικά και για τα γενώσιμα. Θέλω λοιπόν να γίνει σχετική συζήτηση για να προχωρήσουμε στις ανάλογες ε, τροπολογίες και επιλογές. Τώρα για τα εκτός συνταχογράφησης φάρμακα, αυτά τα οποία ονομάζουμε over the counter, εδώ προτείνω να γίνεται αποτίμηση και αξιολόγηση ένα πενταετία από τη στιγμή θέση σε ισχύ δηλαδή της οδηγίας, ώστε να αντιληφθούμε τι είδους μέτρα ασφαλείας θα είναι τα πλέον χρήσιμα. Η πρόθεσή μου λοιπόν με τη διάκριση αυτή και τις διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων που έχω προβλέψει είναι η πρότασή μας να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο λογική και αμέσως να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν, στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μας λείπουν δεδομένα και στοιχεία. Αλλά μέσω αυτών που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας πρέπει να δράσουμε αμέσως. Τέταρτη παρατήρηση τώρα, και εδώ πραγματικά στέκομαι μόνο στα βασικότερα, στις προσθήκες που κάνω στην πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα μέσω του ίντερνετ γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο είναι, μια από τις βασικές διόδους των ε, ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά και γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους εμπορία είναι νόμιμη σε κάποια κράτη-μέλη και σε κάποια άλλη παράνομη. Μου φαίνεται λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ε, τομέα ότι, όπου η ρύθμιση πρέπει να αποσαφινιστεί, πρέπει να διοργανωθεί καλύτερα. Νομίζω ότι δεν θα ήταν απλό να δικαιολογήσουμε στην κοινή γνώμη ότι προτιθέμεθα να μονοθετήσουμε για την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα διανομής και αφήνουμε εκτός τη βασική τους δίωδο, δηλαδή το διαδίκτυο και την πώλησή τους στο ίντερνετ. Θα ήταν δύσκολο να το καταλάβει αυτό η κοινή γνώμη και δύσκολο να το δικαιολογήσουμε και στην προοπτική της διασφάλισης της υγείας των ασθενών. Εδώ παρουσιάζω λοιπόν ένα σύνολο προτάσεων και τροπολογιών συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου με την βασική προτεραιότητα να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού του κινδύνους αγοράς φαρμάκων μέσω ιστοθέσεων στο διαδίκτυο και να ενισχύσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να επιτρέπουν την ευαισθητοποίηση ακριβώ των καταναλωτών ιδίως σε ό,τι αφορά την ύπαρξη παραποιημένων ψευδεπίγραφων φαρμάκων και τους κινδύνους που ενέχει η αγορά των φαρμάκων αυτών μέσω μη νομίμων οδών. Επίσης, προτεραιότητά μας είναι όλοι οι ασθενείς να γνωρίζουν τους ιστοτόπους που υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία και αυτούς που είναι εκτός. Ποιοι δηλαδή σέβονται τα μέτρα που προβλέπει η οδηγία και ποιοι όχι. Στην περίπτωση του Ενωμένου Βασιλείου, εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα τέτοια περίπτωση, διότι υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωσης μέσω του Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, του Βρετανικού δηλαδή φαρμακευτικού οργανισμού, όπου δίνονται σαφείς και πλήρες πληροφορίες για πολλά από αυτά τα στοιχεία. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν πολύ καλά τις τροπολογίες που έχω Υποβάλλει εδώ, αλλά δίνω ένα παράδειγμα απλώς του συστήματος. Μπορεί κανείς να συνδεθεί μέσω των φαρμακεί, μάλλον μέσω του στοτόπου να δει ποια φαρμακή απολούν φάρμακα ή όχι. Και να έχει έτσι γνώση του ποια είναι τα φάρμακα που νομίμως πολλούνται και πού. Εδώ να διευκρινίσω ότι νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να περιληφθεί οπωσδήποτε στην οδηγία αυτό του διαδικτύου. Τώρα για να μην πλατιάσω και να αφήσω και χρόνο για την όλη συζήτηση, εδώ θεωρούμε ότι η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί κλιματική πράξη διότι θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, οπότε πρέπει να ορίσουμε και ποινές για μια τέτοια εγκληματική πράξη, ανάλογες με αυτές που εφαρμόζονται για άλλες παράνομες ενέργειες, όπως αυτές που έχουν να κάνουν με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και αυτό είναι δική μας προσθήκη και διευκρίνηση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Έκτο σημείο τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να δούμε τις καλές πρακτικές παρασκευής, όπως ορίζονται από τις Διεθνείς Συμφωνίες Παρασκευής των Φαρμάκων, και θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι επιθεωρήσεις, οι συνηθισμένες επιθεωρήσεις, αρκετές φορές μας έχουν οδηγήσει στην αντοπισμό ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Όμω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μελέτε κινδύνου στοχευμένε που με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό να βασίζονται στα κριτήρια και τους στόχους του έκτου προγράμματος συνεργασίας, διεθνούς συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή καταργεί τα σύνορα για αυτού του είδου τι επιθεωρήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, διότι όσο πιο ενισχυμένη είναι η διεθνή συνεργασία, τόσο περισσότερο αναπτύσσονται πολυμερείς μηχανισμοί κατάλληλοι ώστε να ενεργοποιούνται οι επιθεωρήσεις και η... και ακολούθως ο εντοπισμός των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και η, εμπειρία τους, η εμπορία τους στην αγορά. Όγδοη παρατήρηση. Το θέμα της ενημέρωσης και των εκθέσεων. Είναι απαραίτητο να δημιουργεί ένα δίκτυο επικοινωνία μεταξύ τη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και των αρμόδιων αρχών του κάθε κράτου μέλου, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα. Είναι υπαρκτό το φαινόμενο αυτό τη διακίνηση ε, ψευδεπίγραφων φαρμάκων και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, διότι όλε οι συζητήσει που έχουμε ω τώρα εδώ είναι θεωρητικέ και πολλέ φορέ μα φέρνουν ε, στο φω και αντιφατικέ πληροφορίε. Δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και πορίσματα. Είναι λοιπόν, λοιπόν σημαντικό τα δεδομένα και τα στοιχεία που υπάρχουν να τα συνδυάσουμε. Και κάποιο να φροντίζει για αυτή την συλλογή των στοιχείων και ετησίω να ε, λαμβάνουμε γνώση του τι διαστάσεις έχει το πρόβλημα και τι δράσεις πρέπει να αναλυθούν. Τελευταία παρατήρηση, εξαγωγές. Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στον έλεγχο και στην διακίνηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων σε τρίτες χώρες και είναι πολύ δύσκολο εδώ να εξηγήσουμε πώς μπορεί να ισχύουν τόσο αυστηρά μέτρα ως προς τους Κανόνε που ισχύουν για τα φάρμακα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση για τα φάρμακα που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Αγορά προ τρίτε χώρε, ιδίω προ την Αφρική και την ε, Λατινική Αμερική ή την Ασία. Το να μην συμπεριληφθεί και αυτή η διάσταση αποδυναμώνει σημαντικά το κύρος της Ευρώπης στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. Πρέπει λοιπόν να υποφεληθούμε αυτή τη ευκαιρία ώστε να ζητήσουμε από τι νομικέ υπηρεσίε να αποσαφηνίσουν πώς γίνεται η κατανομή αρμοδιτήτων στον τομέα αυτό και βάσει της νέας συνθήκης της Λισαβόνας. Σίγουρα κάποια άρθρα της οδηγίας θα πρέπει να αλλάξουν βάσει των, υποχρεώσεων, των νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν. Και τέλος, να πούμε, και αυτό είναι το πραγματικό τέλος, να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει προστιθέμενη αξία στο όλο εγχείρημα, ιδίως ε, στην προσοχή μας συνεργασία. Θα ευχαριστήσω εδώ τους συναδέλφους ειδικότερα, τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Και επειδή αυτή είναι η πρώτη έκθεση που υποβάλλω στο Ευρωκοινοβούλιο, Αναμένω τις ε, τροπολογίες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Είμαι απολύτως στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε επικοδομητικά και για να οδηγηθούμε σε μια τοποθέτηση που θα εκφράζει ως δυνατόν περισσότερο όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μαρίζα Ματίας για την παρουσία στην έκθεση και την τόσο εντατική σας ενασχόληση με τη ε, η υπόθεση αυτή. πρώτη έκθεση και είναι τόσο μεγάλο επίβολο σχέδιο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχουμε τώρα τους σχεώδεις συγητές που ζητούν το λόγο. Η Ντάγμα Ροντ πρώτη. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Μαρίσα Ματίας πραγματικά από την αρχή πήρε ένα θέμα που την έριξε στα βαθιά νερά και έκανε ως καταπληκτική έκθεση θα πρέπει να επενέσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Να είναι από την αρχή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλή. Είναι πολύ καλή και βεβαίως χωρούν και βελτιώσεις και, λείπουν και κάποιοι τομείς, τα είπε η Μαρίσα. Να πω κι εγώ μερικά πράγματα με χαρά. Ποια ε, είναι η κεντρική ιδέα. Ασφάλεια των ασθενών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Η ασφάλεια των ασθενών για μένα ακριβώς ανάγεται στο πού υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος. Γι' αυτό συμφωνώ με τη Μαρίσα Ματίας ότι κατά κύριο λόγο εδώ μιλάμε για συνταχογραφούμενα φάρμακα. Ε, μπορεί να είναι γενώσιμα, ε, κοινόχ της ε, ονομασίας ή ιδιοσκευάσματα. Όταν λοιπόν έχουμε ένα φάρμακο που δεν μπορεί να το αγοράσει κανεί ελεύθερο, αλλά χρειάζεται υποχρεωτική συνταγή, ε, είναι κάτι διαφορετικό από κάτι που μπορώ εγώ να πάρω μόνη μου, γιατί με πονάει το κεφάλι μου. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ορίζεται από το αν είναι υποχρεωτική συνταγογράφηση ή όχι. Η διαφορά δεν είναι και δεν μα ενδιαφέρει αν είναι ιδιοσκεύασμα ή αν έχει δίπλωμα ευρεσιτεχνία ή είναι γενώσιμο το φάρμακο. Και συμφωνώ με τη Μαρίσα, προβλέπει μια πενταετή περίοδο για να δούμε αν θα μπουν και τα φάρμακα γενικά που μπορεί κανείς να αγοράζει ελεύθερα στο φαρμακείο. Over the counter λέγεται αυτό στα αγγλικά. Να δούμε αν θα χρειαστούν βελτιώσεις και συμφωνώ πάντως μαζί ε, καταρχήν να το αναφέρουμε έτσι. Μετά, είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και θα πρέπει να ε, είναι ε, πολύ σημαντικό και ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά όλα δεν είναι ακριβά. Αυτό που μας κοστίζει είναι η, χνηλασιμότητα και η παρακολούθηση. Ε, μα και η ασφάλεια έχει το τίμημά της και θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Προηγουμένως μιλούσαμε για την φαρμακοεπαγρύπνηση και ήταν για μας προφανές και αυτονόητο. επιθύμητες ενέργειες να είναι γνωστές. Ε, εδώ ακόμα περισσότερο. Όταν ένα φάρμακο είναι ε, απειλή, ε, κίνδυνος ή ε, αν δεν έχει ενεργή δραστική ουσία. Ιδιαίτερα για φάρμακα που καταπολεμούν τον καρκίνο ή ρίχνουν την χολυστερόλη. Γιατί αν είναι το φάρμακο χωρίς δραστική ουσία είναι επικίνδυνο γιατί δεν μπορεί να προστατεύσει τη ζωή. θα πρέπει ειλικρινά να συζητάμε τα προβλήματα, γιατί τα βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν οι παράλληλοι έμποροι. Ε, δεν ξέρω ότι θέλει να απαγορεύσει η κυρία Κροστέτος προς τις συσκευασίε στο overboxing. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας να είναι παντού τα ίδια δεδομένα. Δεν ξέρω θα μπει σε αυτή την νομοθεσία ή αλλού. Θέλω να απαγορεύσουμε ε, να κόβονται τα μπλίστερ. Αυτό δεν ασφαλεία για τον καταναλωτή. Ε, τότε είπε ο κύριος ε, Λίζε να είναι ενιαίες οι συσκευασίε και να περιέχουν τον ίδιο αριθμό δισκείων, ας πούμε. Ε, εντάξει, θα δούμε και εκπρόσωποι που έχουν τα συμφέροντά τους, πώς θα υπερασπίζονται και πώς θα προωθούν. Θέλω να πω κάτι τώρα για το βασικό πρόβλημα, που είναι η διάθεση μέσω ε, φαρμακείων στο ίντερνετ. Μας ξεπερνούν οι εξέλιξει. Πριν από πολλά χρόνια ορισμένοι το λέγαμε ότι τα φαρμακεία στο διαδίκτυο είναι κακό πράγμα για τους ασθενείς, διότι καταργείται η άμεση επαφή με τον ασθενή που μπορεί να έχει τα προβλήματά του ή τις ε, έννοιες του, ε, που είχε προσωπική επαφή με το φαρμακοποιό. Αυτό καταργείται. Αλλά στο παρελθόν μας είπανε ε, ότι α, είναι αυτά τα πράγματα, είναι πιο φτηνό, δεν πειράζει. Ορίστε, τώρα ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση. Πολλούνται φάρμακα στο διαδίκτυο. Το είπε και η κυρία Ματίας προηγουμένως. Και να πιστοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, τις ιστοσελίδε τους. Να γνωρίζουν οι καταναλωτές, οι ασθενεί, ποια είναι πιστοποιημένη, εγκεκριμένη ε, σελίδα, ένα εγκεκριμένο φαρμακείο στο διαδίκτυο ε, και αυτό σημαίνει και δυνατότητα αποζημίωσης. Είναι σημαντικό αυτό. Κάτι άλλο που πιστεύω είναι, αν δούμε τα χαρακτηριστικά αυτά ασφαλείας, ότι βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εχνηλασιμότητας. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αν γνωρίζουμε ότι μια παρτίδα ε, δεν έχει δραστική ουσία, είναι εικονικό φάρμακο και το έχει πάρει η Dagmar Rothbard, να της το πούμε επιγόντως ότι είναι ανενεργό το φάρμακο. Και κάποιοι φωνάζουν και ορίονται ότι αυτό φτιάχνει το γυάλινο ασθενή, δηλαδή δεν προστατεύονται τα δεδομένα του και είναι δημόσια αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ε, χάρτης υγείας, ε, η, η ασφάλεια συγγνώμη, των ασθενών είναι πολύ πιο σημαντικό και αυτό που θέλουμε ε, είναι να το προστατεύουμε για να τον βρούμε, να τον ενημερώνουμε, να τον προειδοποιούμε. Αυτά είναι σημαντικά για μένα ζητήματα και στο μέλλον θα εξακολουθούν. Τώρα, σε κάτι που πρότεινε η κυρία Ματίας, έχω επιφυλάξεις για τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις που είναι στις τροπολογίες 12, 24, 25, 37, 45 κλπ. Δεν με έχει πείσει ακριβώς για το πώς θα λειτουργήσει, ομολογώ, και πώς θα γίνεται σωστά ο έλεγχος και ποιος θα τα πληρώνει. Η τροπολογία 42 κακή δεν είναι, αλλά δεν μπορώ να τη φανταστώ στην πράξη. Γνωρίζουμε ήδη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και επιθεωρητές και ελεγχτέ εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ανταποκρίνονται στο πρόβλημα κάτι που πρέπει να εξασφαλίσουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι παρασκευαστές, είτε είναι ίδιο σκεύασμα είτε είναι σκεύασμα γενώσιμο, να έχει εσωτερικό έλεγχο στην εταιρεία που το παράγει να είναι καλύτερος έλεγχος της δραστικής ουσίας και το σκεύασμα αυτό ε, να, να είναι εξαιρετικής ποιότητας. Έχουμε και άλλα θέματα, διαφορετικές ε, κατηγορίες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Εκεί διαφέρω λίγο ίσως με τη Μαρίζα. Στην τροπολογία 9, τουλάχιστον δεν το κατάλαβα πάρα πολύ καλά, μιλάει για διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, ε, διαφορετικά προϊόντα. Δεν το κατάλαβα εκ πρώτης όψεως αυτό. Μήπως είναι υπερβολικά φιλόδοξο και λεπτομέρεια για την αρχή. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Ευχαριστώ. Yeah, σε ευχαριστώ. Και το παράλληλο εμπόριο ήταν συχνά στο χαστρό. Όποιος μπορεί να ανοίξει ένα πακέτο με ένα ψαλίδι μπορεί και να παραποιήσει ένα φάρμακο. Γνωρίζουμε πάντως τώρα ότι οι πηγές του παραποιημένου φαρμάκου είναι αλλού. Γνωρίζουμε τώρα ότι από το παράλληλο εμπόριο τα πράγματα είναι διαφορετικά και ίσως δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε τώρα τα πράγματα. Ας μην ανακατεύουμε τα μεγέθη των πακέτων των φαρμάκων και τα ίδια τα φάρμακα που βρίσκονται μέσα. Η Όλγα Ο, συγγνώμη, ο Χόλγερ Κράμερ. σκιώδη Δεν θα μακρηγορήσω γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ συμφωνούμε για το εάν και πώ θα προωθήσουμε το θέμα. Προπενταετία και εγώ βρισκόμουν στην ίδια θέση μαζί σα. Μόλι μόλις είχα γίνει Ευρωβουλευτή και μου ανέθεσαν μια έκθεση και κολύμψε στα βαθιά νερά. Συγχαρητήρια λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε το θέμα. Υπάρχουν ορισμένα ε, θέματα συστημικού χαρακτήρα, πούμε, όπου έχω κάποια ερωτηματικά. Νομίζω ότι όμως μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Δεν θα επαναλάβω ότι υπάρχει κίνδυνος παραποίησης φαρμάκων και στην Ευρώπη, είναι σαφές αυτό. Ένα πράγμα που δεν κατάλαβα πολύ καλά είναι για ποιο λόγο η συγγήτρια γιατί ε, θέτει το θέμα των εκδόχων. Στο νομοθετικό κείμενο πάμε με τον τρόπο αυτό να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής και στην παραγωγή των φαρμάκων. Ενώ από όσο ξέρω υπάρχουν επαρκείς νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα αυτό και διαρωτώ με αν όντως εξυπηρετεί τον σκοπό μας εάν πάμε να κάνουμε ακόμα πιο αυστηρές τις ήδη αυστηρές προδιαγραφές για την παρασκευή των φαρμάκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι την προσοχή μας πρέπει να, να δώσουμε κυρίως στην διακίνηση των φαρμάκων. Δεν είμαι λοιπόν σίγουρος ότι αυτό το συγκεκριμένο μας εξυπηρετεί. Και η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, είναι αρκετά σαφής με την συμπλήρωση ορισμένων διατυπώσεων για τα generics έχω την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται περισσότερο να τα αποκλείσουν από τη διαδικασία αυτή αντί να τα περιλάβουν. Τουλάχιστον αυτό κατανοώ από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σωστό θα ήταν να βασιστούμε στον ενδεχόμενο κίνδυνο και να δούμε σε ποια από τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται χωρί συνταγή, υπάρχουν ενδεχομένω κίνδυνοι και όπου πρέπει να μπουν κάποια χαρακτηριστικά ασφαλεία. Δεν μου φαίνεται σκόπιμο τα φάρμακα χωρί ειδική επωνυμία, τα generics, να χρειάζεται να ε, γίνει κάποια συγκεκριμένη άλλη ε, πρόβλεψη για αυτά. Γιατί θα έχουμε και ε, από τη μια μεριά θα έχουμε τα φάρμακα με επωνυμία τα οποία, για τα οποία δεν απειλείται να υπάρξει παραπίση και θα έχουμε τα generics όπου μπορεί να υπάρχει παραπίση. Για το διαδίκτυο, σωστό μου φαίνεται αυτό που γράφεται και η κυρία Ροτ Πέρεντ ίσως ορισμένα πνεύματα εντό εισαγωγικών να μην χρειάζεται να τα καλέσουμε ειδικά, εμφανίζονται από μόνα τους. Δεν θα μπορέσουμε να παρεμποδίσουμε δηλαδή να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία το διαδίκτυο και ο ασθενής ο οποίος παραγγέλνει φάρμακα με το διαδίκτυο και τα λαμβάνει πρέπει να γνωρίζει ότι διατρέχει έναν κίνδυνο. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να τονίσουμε τους κινδύνους του διαδικτύου. Τώρα, πιστοποιημένα φάρμακα, τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση, αν θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος ετικέτα, ένα label του διαδικτύου. Πάλι και αυτό μπορεί να παραποιηθεί και αυτό είναι σαφές. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Κάτι που μου φαίνεται υπερβολικό είναι η ιδέα να ε, υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει φραγμούς μέσα στα λεγόμενα search engines του διαδικτύου. Τις ε, μηχανές αναζήτησης δηλαδή. Αυτά είναι τα σημεία όπου θεωρώ ότι χρειάζεται να τα ψάξουμε λίγο ακόμα. Κατά τα άλλα, η γνώμη της ομάδας μου είναι θετική και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη. Äh, Απούσα. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την ε, κυρία Μαρίζα Ματίας, για την ε, εξαιρετική και εμπεριστατωμένη εισήγηση που έκανε. Έχει καλύψει σε έκταση το θέμα και αρκετά από τα ζητήματα που θέλαμε να τονίσουμε τα περιέλαβε και έκανε τη δουλειά μας πιο εύκολη. Οι περισσότερες ε, τροπολογίες της καλύπτουν τα βασικά αιτήματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ε, σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο και μας βρίσκουν σύμφωνος. Θα πρέπει να επιμείνουμε όμως σε κάποια σημεία ιδιαίτερα. Καταρχάς, η επιχειρηματολογία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αναλωθεί σε συζητήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και το παράλληλο εμπόριο ή ακόμα και τα αντίγραφα φάρμακα, καθώς αυτά αφορούν κυρίως εμπορικές διαστάσεις και όχι τόσο την προάσπιση του δημόσιου, του συλλογικού συμφέροντος και της, ε, συλλογική, της δημόσιας υγείας. Ε, και στο προήμερο αλλά και στους ορισμούς η κυρία Ματίας μας καλύπτει διαχωρίζοντας τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και των πατέντων. Δεύτερον, πρέπει να εισάγουμε ρυθμίσεις για να καταπολεμήσουμε όντως τις παράνομες διαδικτυακές πωλήσει, την κύρια πηγή των ε, ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Η πρόταση της Επιτροπής ασχολείται με την ε, παραδοσιακή αλυσίδα διανομής ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά, ενώ όπως γνωρίζουμε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για να καταπολεμήσουμε τις ε, παράνομες διαδικτυακές πωλήσει. Υπάρχουν κάποιες ιδέες έστω και αν από νομική σκοπιά η οδηγία δεν μπορεί να εισαγάγει άμεσες ρυθμίσεις για διαδικτυακά φαρμακεία και παράνομες πωλήσει. Οι προτάσεις της κυρίας Ματίας, οι τροπολογίες συγκεκριμένα από 39 έως 41, για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού μητρώου πιστοποιημένων διαδικτυακών φαρμάκων, φαρμακείων σε χώρες όπου επιτρέπεται η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων καθώς και δημιουργία ενιαίου λογοτύπου πιστοποίησης διαδικτυακών φαρμακείων είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να έχουν πιο συστηματική συνεργασία και μέσω της Europol για να εφαρμόσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την αποτροπή των παράνομων πωλήσεων μέσω του διαδικτύου και, ότι, και το ότι αυτή η οδηγία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπονομεύσει το δικαίωμα των κρατών μελών να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την αγορά των ε, συνταγογραφημένων φαρμάκων από το διαδίκτυο. Τρίτο σημείο, πρέπει να υπάρχει ένας πιο ξεκάθαρος ορισμός για το τι είναι ψευδεπίγραφο φάρμακό με βάση τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μόλις του Δεκεμβρίου του 2008, ούτως ώστε να διατηρήσουμε συμπαγή τη διεθνή συνεργασία των κρατών μελών. Ο ορισμός της ε, κυρίας Ματίας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τέταρτον, χαιρετίζω την πρόθεση της Επιτροπής για ενδυνάμωση των ελέγχων όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διανομής, όπως επίσης και όλων των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών. Θα ήθελα να μεταφέρω το αίτημα για υποχρεωτική εγγραφή σε Μητρό όλων των εμπλεκομένων στην ομοια αλυσίδα παραγωγής διανομής, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό. Μας ικανοποιεί που γίνεται η αναφορά σε πιο αυστηρούς ελέγχου από την κυρία Ματίας στι τροπολογιε 42 42-43, αλλά και απόδοση ποινικών ευθυνών και όχι μόνο προστήμων. Πέμπτο σημείο. Θεωρούμε σημαντικό που γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ότι ε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εξαγωγή και διανομή πιστοποιημένων φαρμάκων σε τρίτες χώρες. Τα άλλα υπόθηκαν. Συμφωνούμε με τις προτάσεις σχετικά με το repackaging, η τροπολογία 30, αρκεί να γίνεται υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών και με τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας. Τέλος, πρέπει να υπάρχει συνεχής και ξεκάθαρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για να κάνει λογικές και υπεύθυνε αγορές καθώς και για να συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό και την αναφορά των παράνομων ενεργειών και φαρμάκων. Οι προτάσεις της ηγήτριας μας βρίσκουν σύμφωνος. Αν και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα επίσης το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κατανοητικέ του συνήθειε. Και κλείνω με ένα σχόλιο στην τροπολογία, στην οποία δεν συμφωνούμε κι εμείς. Είναι η 28, καθώς θεωρούμε ότι όλα τα φάρμακα που συνταγογραφούνται, συμπεριλαμβανομένων των generics, πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας. Σε άλλη περίπτωση, η προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα φάρμακα που συνταγογραφούνται, ούτως ώστε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας να ισχύουν για όλα. Σας ευχαριστώ. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλούς ακόμη παρεμβαίνοντες έχω. Οι επόμενοι θα πρέπει να μιλήσουν από δύο λεπτά ο καθένας, Η δεν θα προλάβουμε. Λίζε, ευχαριστώ. Μια σύντομη προκαταρκτική παρατήρηση πρώτα να πω ότι η κυρία Γκροστέτ κολλείεται και ίσως μου επιτρέψετε να τα πω εγώ κάνοντας μια εξαίρεση που είναι η ίτρια δηλαδή της ε, πολιτικής ομάδας του Λαϊκού Κόμματος. Ε, αν δεν μου το επιτρέψετε αυτό να μιλήσω για λογαριασμό της δηλαδή θα μιλήσω εγώ μόνο για τα δύο δικά μου λεπτά. Η κυρία Κροστέτ, λοιπόν είχε σημαντική αντιλημμένη υποχρέωση. Εμένα μου τα έθεσαν υπόψη την τελευταία στιγμή τα πράγματα αυτά. Στην ομάδα εργασίας μας βέβαια κάναμε μια συζήτηση και μπορώ να σας πω περίπου τι σκέπτεται κυρία Γροσέτα αλλά και όλη η πολιτική ομάδα του Λαϊκού Κόμματος. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι καλή η έκθεση της κυρίας Ματίας, ότι αποτελεί καλή βάση για την εργασία μας και υποστηρίζουμε καταρχήν τις προτάσεις της. Ιδίω η κυρία Γκροστέτ αναφέρεται στην διπλή νομική βάση και είμαστε υπέρ υποστηρίζουμε ακόμη την ανάγκη ενός ακριβέστερου ορισμού ότι δεν πρόκειται για πειρατεία προϊόντων, σημαντικό θέμα αυτό βέβαια, ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι το ότι πρόκειται περί φαρμάκων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν και σημαντικές βλάβες. Γι' αυτό χρειάζεται ένας ακριβέστερος ορισμός. Το υποστηρίζει και η Αγκοστέτ και εμείς. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, εφαρμογής της οδηγίας, κυρώσεις, τροπολογίες 13 και 14 μας βρίσκουν σύμφωνους και βέβαια και οι τροπολογίες για την διάθεση μέσω ίντερνετ. Η κυρία Κροστέτ λέει ότι ίσως στην μεταβατική περίοδο θα έπρεπε να την προβλέψουμε συντομότερη. Η κυρία Σαρτόρη στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών πρότεινε θέση σε εφαρμογή μετά από εξάμεινο. Ίσως αυτό είναι υπερφιλόδοξο. Ίσως μπορεί να προκύψει ένα συμβιβασμό. Και στο θέμα αυτό να τα βρούμε περίπου στη μέση με την ΙΜΚΟ. Βέβαια, όπως είπε και η κυρία Ροτ Μπέρεντ, υπάρχει και η πρόταση της κυρίας Γκροστέτ για το λεγόμενο overboxing, δηλαδή μια γενική απαγόρευση ανοίγματο των συσκευασιών. Μεταφέρω την ιδέα αυτή, κλείνω τα σχόλια της κυρίας Γκροστέτ. Βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Εγώ προσωπικά μπαίνω στο δεύτερο μέρος τώρα της παρέμβασής μου. Έχω κάπως κριτική στάση απέναντι στο λεγόμενο overboxing γιατί δεν έχουμε ακόμα ενία μεγέθη συσκευασιών και ούτε νομίζω θα μας προκύψουν και γρήγορα. Και γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για, τον, για την πώληση μέσω ίντερνετ, συμφωνώ με τους προαλήσαντες συναδέλφους, προσθέτω το εξής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δίνει στις χώρες μέλη την δυνατότητα να απαγορεύσουν γενικά την πώληση μέσω ίντερνετ για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο μετά από συνταγή. Οπότε θα μπορούσαμε έτσι να κλείσουμε το κενό. Τελευταίο μου σημείο είναι ότι θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια για την ίχνη λασιμότητα να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Όσα είπε η κυρία Ροτμπέρεντ είναι σωστό. Εάν κρυθεί κάποιο φάρμακο παραποιημένο πρέπει να ειδοποιείται ο ασθενής. Υπάρχει όμως και ο δικαιολογημένος φόβος ότι ενδεχομένως ένας παρασκευαστής φαρμάκων μπορεί και να καταχραστεί αυτής της πληροφορίας εάν γνωρίζει δηλαδή ποιοι γιατροί συνταγογραφούν ποια φάρμακα και ποια ε, φαρμακεία πολλούν ποια φάρμακα κτλ. μπορεί να γίνει κατάθεση των πληροφοριών αυτών. Άρα χρειάζεται ειδική προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Ω, τηρήσατε, τηρήσατε ακριβώς τον χρόνο σας, δύο λεπτά για την κυρία Γκροστέτ και δύο, λεπτά για εσάς. Η κυρία Πραβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, θα χρειαστεί ε, να πείτε πολλές φορές το όνομά μου φαίνεται και θεωρήστε το αυτοπρόσκληση σε καφέ μέχρι να το μάθετε. Πολύ καλή δουλειά η Ματίας έκανε για τη νομική βάση κυρίως και για την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων το διαδίκτυο και την ενίσχυση της συνεργασίας ε, για ε, την εκπαίδευση των τελωνιακών. Έχω τα εξή σημεία να σας ε, θέσω υπόψη. Όταν συζητούμε για το διαδίκτυο, το θέμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το διαδίκτυο που πολύ το προϊόν. Θα περάσει και από ένα τελωνίο μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Να σας δώσω ένα αστείο ίσως παράδειγμα, αλλά έχω τους λόγους μου. Προσπαθήστε να στείλετε με τη DHL ή τη FedEx χρήματα από πιστοτική κάρτα. Δεν πρόκειται να το καταφέρετε για τον εξή καλό λόγο. και για εύλογου λόγου. Ανοίξαμε την πόρτα, πουλάμε πολύ επικίνδυνα προϊόντα όπω είναι τα φάρμακα μέσω του διαδικτύου και ε, τώρα έχουμε μπλέξει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θα πρέπει να καταλάβουν οι καταναλωτές, να τους ευαισθητοποιήσουμε τους ασθενείς να αγοράζουν φάρμακα όχι από το φαρμακείο της γειτονιάς τους ή κάποιο πιο μακριά, αλλά από ένα εικονικό φαρμακείο, διαδικτυακό. Ε, για τα διασκευάσματα, για τα γενώσιμα φάρμακα. Ή τα over the counter που δεν χρειάζονται συνταγή. Αν τα εξαιρέσουμε αυτά, τα γενώσιμα φάρμακα δεν ε, αντιγράφονται τόσο πολύ. Είναι λιγότερο το τα OTC αντιγράφονται περισσότερο. Είτε θα τα βάλουμε και αυτά, είτε θα βγάλουμε και τα γενώσιμα, γιατί τελικά τα... θα καταντήσει ένα ε, φάρμακο που κάνει 3 ευρώ να κάνει 4 ευρώ. Και θα πρέπει και η τιμή να είναι ένα στοιχείο. Και το τελευταίο, η επανασυσκευασία. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό Δηλαδή, ως προς το χρονοδιάγραμμα, η νομοθεσία μας δεν πρόκειται να ε, εκδοθεί, να τεθεί σε ισχύ πριν την επόμενη τριετία και θα συνεχίζουν τα κράτη-μέλη να ε, εφαρμόζουν τη δική τους νομοθεσία για τη συσκευασία. Δεν έχω δει πουθενά κανένα προϊόν που να κυκλοφορεί στην Ευρώπη να το ξανασυσκευάζουν. Ρώτησα, υπάρχουν τέτοια προϊόντα. Μου λένε αυτοκίνητα. Δηλαδή τι τα κάνουν, τα, τα, τα ανοίγουν και μετά τα ξανααμπαλάρουν. <clears throat> Μόνο στα φάρμακα συμβαίνει αυτό και είναι πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Παρβάνοβα, σας είπα τώρα σωστά, το πέτυχα. Και σα ευχαριστώ και την πρόσκληση για καφέ. Γιάννα Σάντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω εδώ μια συνήθιστη μέθοδο και ζητώ την άδειά σας. Να κάνω ερώτηση στην εισηγήτρια μου επιτρέπετε και στους σκιώδεις εισηγητές και μετά την απάντηση να μου ξαναδώσετε το λόγο, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ρωτήστε. Δεν έχουμε χρόνο. ρωτήστε, αλλά θα σας απαντήσει στο τέλος η συγκήτρια. Αλλιώς δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, εγώ περίμενα η απάντηση να είναι μία λέξη ή ένας αριθμός. Δεν θα μας έτρωγε και πάρα πολύ χρόνο. Εν πάση περιπτώσει. Έχω την εξής ερώτηση να κάνω. Γνωρίζει κανένας από τους παρόντες εδώ το ποσοστό των ψευδεπίγραφων φαρμάκων που πολλούνται στο διαδίκτυο. Εγώ το συζήτησα με διάφορους εμπειρογνώμονες και δηλώνουν ότι είναι 80 με 90%. Ξέρω όμως και άλλα νούμερα που ακούγονται. Ε, πάντως είναι γεγονός ότι τα μισά και πλέον ψευδεπίγραφα, των φαρμάκων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι ε, Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή. Η κυρία Ματίας είπε ότι στο αρχικό κείμενο ε, ε υπήρχε μια τέτοια ένδειξη και ο κύριος Φερχόιγκεν είχε πει ότι στην αρχή έγιναν πολλές κατασχέσεις δισκίων και φαρμάκων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λέει ούτε λέξη για την πώληση στο διαδικτύο. Ενώ η συγγήτρια θέλει να τα συμπεριλάβει. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα έτσι. Εγώ από αλλού περιμένω λύση. Το ανέφερε και αυτό η συγκήτρια. Δηλαδή, να επιστήσουμε την προσοχή των κρατών μελών στο εξή γεγονός. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να απαγορεύσουν τα ηλεκτρονικά φαρμακεία στο διαδίκτυο, γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιούντιτ ε, Μέρκης. Uh, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Ματίας για μια έκθεση πολύ τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη και με μια καλή αντίληψη για το τι συμβαίνει στη βιομηχανία και στο επίπεδο των καταναλωτών. Εδώ νομίζω ότι την υγεία των ασθενών πρέπει να την έχουμε ω πρώτη προτεραιότητα. Αυτό είναι σαφές. Όμω, πρέπει να τονίσω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πρόταση κατά των παραποιημένων φαρμάκων. Αυτό θα πρέπει να έχουμε συνεχώ κατά νου. Πράγματι, είναι σημαντικό ότι έχουμε συμπεριλάβει και τις καταχρήσεις της αγοράς στο διαδίκτυο και θα, θα συμφωνήσω με την κυρία Ντάγμα Ροτέρεντ ότι πρέπει να είναι ασφαλείς και οι πηγές μας, αλλά επίσης σημαντικό είναι να ενημερώνεται και ο καταναλωτής για τον κατάλογο με τις ασφαλείς πηγές που θα έχουμε καταρτήσει εμείς, για να ξέρει και πώς θα τον χρησιμοποιήσει. Ιδάλλως δεν έχει νόημα να έχουμε ένα κατάλογο με τις ασφαλείς πηγές μόνο εμείς στη διάθεσή μας. Επίση, πρέπει να έχουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ε, φαρμάκων που συνταγογραφούνται και αυτών που δεν συνταγογραφούνται <clears throat> και μόνο τα συνταγογραφούμενα θα πρέπει να καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό. Ήδη αναφέρθηκε ότι ο ορισμός των ψευδεπίγραφων και των over the counter βάσει του ορισμού του ΠΟΗ είναι ορισμοί που πρέπει να συνοδευτούν από τα σφάλματα, τα ηθελημένα και τα σφάλματα παρασκευής. Και τελευταίε δύο παρατηρήσει της κυρία Ματίας με τι οποίε δεν συμφωνώ πλήρω είναι οι τακτικέ επιθεωρήσεις και γενικότερα επιθεωρήσεις και ο έλεγχο. Πρέπει εδώ να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν μπορούμε να επιθεωρήσουμε όλο τον κόσμο και να είμαστε βέβαιοι ότι τίποτε δεν θα περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορούμε όμως να ενισχύσουμε το υπάρχον σύστημα, το σύστημα επιθεωρήσεων δηλαδή, όπου θα καλούμε τους παρασκευαστές και θα απευθυνόμαστε στη δική τους ευθύνη να επιθεωρούν την, τα προϊόντα τους και την πηγή τους. Ο κύριος Ναι, ξέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι σημαντικό. Όμως δεν πρέπει να περιορίσουμε τις προσπάθειές μας στην καταπολέμησή του. Ούτε μπορούμε να εμποδίσουμε την πρόσβαση των τρίτων χωρών σε φάρμακα όπως τα γενώσιμα, διότι πέρσι ήδη είχαμε πολύ σημαντικές αποφάσεις με ε, σημαντικές συνέπειες για χώρες όπως η Βραζιλία και άλλες. Μιλάμε λοιπόν εδώ για παραποιημένα φάρμακα που κάποιες φορές δεν είναι καν παραποιημένα. Εδώ λοιπόν πρέπει να ε, πω στην εισηγήτρια ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο με τη δουλειά σα. Ε, κάνατε πολύ καλή δουλειά σίγουρα, αλλά η τροπολογία 3 με δυσκολεύει λίγο, διότι λέτε ότι δεν πρέπει να επηρεαστεί εδώ η νομοθεσία μα. Τα δύο ζητήματα όμω δεν μπορούν να επηρεαστούν το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών. Εδώ σίγουρα θα επηρεαστεί, γιατί κάποια φάρμακα είναι πολύ ακριβά. Οπότε η λογική είναι ότι θα υπάρχει μεγάλο κέρδο. Και αυτό θα σκεφτεί κανείς και θα βάλει σκοπό. Εάν αναθεωρήσουμε το σύστημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών για τα αντιβιωτικά, τα εμβόλια και θέλουμε να προωθήσουμε την έρευνα σχετικά, και αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση των, του κέρδους βάσει της τιμής, Σίγουρα κανεί θα έχει απολαυέ ανάλογα με την έρευνα που έχει κάνει και το προϊόν που θα πουλήσει. Όμω ο κάθε παρασκευαστή θα θέλει να κατασκευάσει το προϊόν μα στο δυνατό μικρότερο κόστο. Οπότε κάποιοι σίγουρα θα παρασκευάσουν ε, τέτοια φάρμακα και θα προσπαθήσουν να τα παραποιήσουν. Δεν θέλω λοιπόν αυτό να εξελιχθεί. Διότι θα πρέπει να δούμε το τι αντίκτυπος υπάρχει στο κόστος παραγωγής και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ίσως και αυτός είναι ένα, ένας τρόπος να εξετάσουμε το σημείο αυτό ώστε να διασφαλίσουμε την καταπολέμηση των ψευδοπλήρων φαρμάκων και από αυτήν την άποψη. Τα ρολόγια στο κοινοβούλιο δείχνουν το καθένα διαφορετική ώρα και κανένα τη σωστή. Μυστήριο για μένα αυτό. Πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέσσερα λεπτά παρακαλώ να λάβει θέση και μετά η άλλα τέσσερα λεπτά ε, και θα τελειώσει ο χρόνο στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τηρήσω το τετράλεπτο και θα είμαι σύντομος. Ωστόσο, θα ήθελα παρόλα αυτά και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Ματίας. Πολύ σύντομα, επί της ουσίας. Πιστεύω ότι τα μέτρα που προτείνονται για το διαδίκτυο είναι σε μια κατεύθυνση που ελπίζω να μην ε, οδηγήσουν σε μια, καμία δυσκολία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην χρειαστεί νομοθεσία για την εναρμόνιση του εμπορίου στο διαδίκτυο. Οπότε υποθέτω ότι δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους θα ήθελα να πω ότι εδώ στο σχέδιο έκθεσης συμπεριλαμβάνεται ένα σημείο που έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις και από πλευράς αξιολόγησης κινδύνου ενδεχομένω να χρειαστεί επανεξέταση. Δηλαδή, ε, ε, τα λεγόμενα έκδοχα που είναι ε, βοηθητικές ουσίες. Είναι διαφορετικός ο κίνδυνος από τη δραστική ουσία που μπορεί να έχει μια τέτοια βοηθητική ουσία του φαρμάκου για να δράσει. Εδώ χρειάζεται προσοχή μάλλον. Τώρα για τις κυρώσεις. καταβάλλονται προσπάθειες στο Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκριθεί η σύμβαση και οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν οριμάσει πολύ, έχουν προχωρήσει πολύ. Και εδώ χρειάζεται προσοχή να μην δημιουργήσουμε ε, ρυθμίσεις δεσμευτικές ε, σε ανταγωνισμό. Τώρα για τον ορισμό των ψευδεπίγραφων φαρμάκων κανένα πρόβλημα και από την αρχή δεν ήταν ε, επίμαχο αυτό το θέμα, ότι νομίζω είναι προβληματικό στη συνέχεια. Το θέμα των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Ναι, και για μένα είναι πρόβλημα να έχουμε διαφορετικά ε, χαρακτηριστικά ε, ασφαλείας για διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων. Θα είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση με μελέτης αντικτύπου και τα λοιπά, για να μην μιλήσω για το κόστος αρμογής. Αν σκεφτεί κανείς και μόνο πόσο δύσκολο είναι σε ένα φαρμακείο σε μια φαρμακαποθήκη να γίνονται ε, επαληθεύσεις για κάθε χαρακτηριστικό ασφαλείας. Το θεωρώ πολύ περίπλοκο αυτό. Και ε, το τελευταίο, για τη θέση ισχύ, βεβαίως θα πρέπει το συντομότερο να τίθεται σε ισχύ όλες οι προδιαγραφές προστασίας, αλλά ίσως να χρειαστεί εδώ μια διάκριση, έτσι ώστε και κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των ελέγχων να επιλέξουμε ένα πιο ρεαλιστικό χρονικό ορίζοντα για να προετοιμαστούν και οι τρίτες χώρες αν έχουμε νέες προδιαγραφές και διατάξεις για τις εισαγωγές. Λοιπόν, όσο και βλέπω και εγώ θετικά ε, το σύντομο χρονοδιάγραμμα να είμαστε κάπως πιο ρεαλίστες. Ε, έχουμε επιθεωρητές του Συμβουλίου της Ευρώπης εν μέρη και των κρατών μελών σε τρίτες χώρες και εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσο οι πόροι ε, που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να πούμε ότι αρκούν για ταχεία βελτίωση. Εμείς προτείναμε να γίνουν έλεγχοι και επιθεωρήσεις, αλλά επιθεωρητές δεν είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Βεβαίως είμαστε υπέρ πιο αυστηρών κανόνων και στις τρίτες χώρες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, αλλά πάντα αναλογικά και ρεαλιστικά. Τελειώσαν τα τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Oh, Ακριβώς επάνω στην ώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Τιλμπεργκερ. Η συγκήτρια έχει τώρα τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συνοδέλφους. Προφανώς σε τέσσερα λεπτά δεν θα προλάβω να απαντήσω <clears throat> στον καθένα ξεχωριστά. Αλλά να εκφράσω εδώ την ικανοποίησή μου για το σύνολο των σχολείων που έγιναν στα σημεία στα οποία είχα και εγώ σταθεί. Νομίζω ότι θα πετύχουμε αρκετά υψηλό βαθμό συμφωνία μεταξύ μας. Άλλα τα σημείωσα μέσα από τη συζήτηση και θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία πρέπει να εμβαθύνουμε, γιατί εδώ το ζήτημα ενέχει πολλούς κινδύνους και στις άλλες αρμόδιες επιτροπέ και με όλες τις συζητήσει που θα γίνουν και με τις τροπολογίες που θα προβληθούν. Είναι σαφές ότι παραμένουν κάποια ζητήματα ανοιχτά, όπως τα χαρακτηριστικά ασφαλεία, safety features, το πεδίο της οδηγίας, τι θα γίνει με τις επιθεωρήσεις. Αυτό θα συζητηθεί σίγουρα ακόμη περισσότερο. Και εδώ θα συζητήσω και διευκρινήσεις για τις αλλαγές που θα επιφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως είχα πει και, την... και προηγουμένως, και σε σχέση με τα άρθρα που θα χρειαστεί να αλλάξουν ως επακόλουθο τις θέσεις σε ισχύ της νέας συνθήκης. Και νομίζω σημαντικό είναι να ακούγονται όλες αυτές οι διαφορετικές θέσεις και να προσπαθήσουμε να τις ε, συνενώσουμε. Το άλλο που θέλω όμω να ρωτήσω οπωσδήποτε είναι τι θα γίνει με τη συμπερίληψη του διαδικτύου και τι άποψη έχει γι' αυτό η Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι από αυτά που σχολιάστηκαν περισσότερα από όλα τα άλλα σημεία και είναι σημαντικό για τις επιθεωρήσεις, για τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν πρόλαβα να έχω μια απάντηση έτοιμη για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν, όμως Πρόεδρε, η Επιτροπή από κοινού με τα κάτι μέλη θα πρέπει να ασχοληθεί σε συντονισμένες προσπάθειες για την επικοινωνία με τις αρχές τρίτων χωρών. Ίσως δεν το αποσαφήνισα καλά στην αρχική μου παρέμβαση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση έχουμε μια καλή βάση για να διαπραγματευτούμε και για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα σημεία που έχουν τεθεί και για τα χαρακτηριστικά ασφαλεία. την ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας και όλα τα άλλα ζητήματα γενικά έχουμε προτάσεις πολύ απλούστερες και πιο εύκολες να εφαρμοστούν από ό,τι προηγουμένως. Και αυτό για την ε, επιδίωξη των στόχων που έχουμε θέσει και παρά την έλλειψη επαρκών δεδομένων. Δεν θα επαναλάβω το ρόλο μου την προηγούμενη παρέμβαση. Απλώ τι μεμονωμένε ενστάσει τι έχω σημειώσει και σαφώ θα συζητήσουμε περαιτέρω για να καταλήξουμε στην επιθυμητή συμφωνία. Ευχαριστώ. Yeah, ε. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 9 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία τον Απρίλιο. Λήξη τη σημερινή συνεδρίαση, αύριο το πρωί στι 9 οι συντονιστές παρακαλώ.